Καλημέρα σας. Έχουμε ούτε το πολλό το F. Έχουμε ποιότητα, όχι ποσότητα. Εξαιρετικά μέλη παρόντα εδώ σήμερα το πρωί για να αρχίσουμε τις εργασίες μας και η πρώτη έκθεση είναι του κυρίου Ντεκάμπος και αφορά τα φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή. Θα συζητήσουμε λοιπόν ε, το 8 και το 9 μαζί. τροποποίηση του κανονισμού και τροποποίηση της οδηγίας. Θα δώσω το λόγο λοιπόν καταρχάς στον κύριο Ντεκάμπο, εν συνεχεία στον κύριο Μπουζόη και εν συνεχεία στους σκιώδεις εισηγητές. και ε, θα ήθελα να συγχαρώ ε, το μέλος μας, το οποίο είναι, είναι το πιο συνεπές ε, όσον αφορά την παρουσία τους εδώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, λέει ο κύριος Ντεκάμπος. Καλημέρα σας συνάδελφοι. Αυτός ο κανονισμός είναι ένας σύντομος κανονισμός, αλλά ε, άπτεται της οδηγίας και γι' αυτό οι επιπτώσεις, ε, οι επιπτώσεις ε, του κανονισμού θα επηρεάσουν ολόκληρη την οδηγία. Το θέμα αφορά έναν ασθενή, μια ασθενή η οποία θέλει να ξέρει τι φάρμακα λαμβάνει για τη θεραπεία της ασθένειάς της. Δηλαδή η πληροφόρηση των καταναλωτών, πώς θα την παράσχω και σε ποιον και ποιος θα τη δώσει το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή δημιουργεί στρεβλώσεις στην ε, εσωτερική αγορά, διότι πολλές φορές οι πληροφορίες αυτές μπορούν να παρασχεθούν σε ορισμένες χώρες, σε άλλες δεν μπορούν λόγω της αυστηρής ερμηνείας, της ε, κυριολεκτικής ερμηνείας ε, της οδηγίας. Αυτή η πληροφορία πρέπει να έχει τρεις πτυχές. Να είναι αξιόπιστη, να βασίζεται στην τρέχουσα επιστημονική γνώση και να είναι ανεξάρτητη, ουδέτερη δηλαδή. Θα πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό μεταξύ του ποιος παρέχει τη χρηματοδότηση, ποιος χρηματοδοτεί αυτή την πληροφόρηση και ε, αν είναι ε, ευνόητη, αν είναι καταληπτή, έτσι ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να καταλάβει τι λέει και να εξασκήσει επίσης μια προσωπική, να, να μπορέσει να διαμορφώσει μια προσωπική άποψη. Να είναι λοιπόν ουδέτερη, ανεξάρτητη αυτή η πληροφόρηση. Αυτό δεν συμβαίνει πολλές φορές. Ε, τα πληροφοριακά ε, δελτία είναι εξαιρετικά περίπλοκα. Πολλές φορές ο γιατός δεν μπορεί να εξηγήσει ακριβώς ε, τη συνταγή την οποία παρέχει στον ασθενή Υπάρχουν βεβαίως πολύ καλές πρακτικές, ε, βέλτιστες πρακτικές ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Σουηδία και στην Πολωνία. Η διαδικασία αυτή είναι πάρα πολύ ικανοποιητική. Αυτή λοιπόν η διαδικασία ενημέρωση δεν θέλει να παρεμποδίσει τη σχέση γιατρού ασθενούς, αλλά έχει ως στόχο να αποσαφηνίσει και να διαφωτίσει και τις δύο πλευρές. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια προκαταρτική εξέταση ε, της, ε, των, ε, της συνταγής και της ενημέρωσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση Φαρμάκων και θα πρέπει η υπηρεσία αυτή να σεβαστεί μία προθεσμία για να παράσει αυτές τις πληροφορίες. Εμείς λέμε 100 20 μέρες προτείνουμε δηλαδή για τα απαντήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση Φαρμάκων όταν τη ζητηθεί γνωμοδότησή της. Όχι 60, 60 πιστεύουμε είναι πολύ σύντομο το, η περίοδος, 120 μέρες. Εάν πιεστεί υπερβολικά χρονικά, τότε μπορεί να παράσχει αντιφατικές πληροφορίες που θα μπερδέψουν ακόμα περισσότερα. Η, η μία, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση Φαρμάκων, θα πρέπει να έχει μια εύλογη προθεσμία για να απαντήσει ε, και να εξετάσει αυτή την παροχή πληροφοριών σε διάφορες γλώσσες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπουρζόη, Κριστιαν Μπουρζόη. Μπουζόη. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πιστεύω ότι οι δύο αυτές προτάσεις για την ενημέρωση των ασθενών, οι δύο αυτές προτάσεις που συζητάμε σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικές και για τις δύο πλευρές, και για τον ασθενή και για ε, τις φαρμακευτικές εταιρείε. Στο Συμβούλιο τώρα ε, έχει επέλθει ένα αδιέξοδο. Πιστεύω όμως και είμαι πεπισμένος ότι αυτή αυτές ε, οι δύο προτάσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές όπως και οι άλλες πτυχές του φαρμακευτικού πακέτου. Και γι' αυτό πρέπει να περάσουν αυτές οι δύο προτάσεις. Τις υποστηρίζω και πιστεύω ότι πρέπει να περάσουν. Η σύνταξη αυτής της ε, ε, πρότασης, αυτής της γνωμοδότησης δεν ήταν καθόλου εύκολη διότι από τη μία πλευρά έπρεπε να εξισορροπήσει τα δικαιώματα των καταναλωτών και από την άλλη να απαγορεύσει την ανάπτυξη των, των, διαφημίσεων των φαρμάκων, των διαφημιστικών εκστρατιών που γίνονται. Επίσης, η άλλη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε είναι διάφορες ερμηνείες ε, για, τις, ε, για τους περιορισμούς ε, παροχής συνταγών στα φάρμακα ή διάφορες κανόνες, διάφοροι κανόνες που μπορούν να ερμηνευθούν ή ευέλικτα ή πάρα πολύ αυστηρά για το αν απαιτείται ή όχι ιατρική συνταγή. Σε μία λοιπόν ενιαία εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέτοιες διαφοροποίησεις και διακοιμάνσεις είναι αρνητικές. Δεν τις θέλουμε στο σχέδιο γνωμοδότησης προτείνω ε, πολλές διευκρινήσεις ε, και αποσαφηνήσεις της αρχικής πρότασης. Οι πληροφορίε, η ενημέρωση αυτή στον καταναλωτή πρέπει να είναι αξιόπιστη και να προέρχεται από αξιόπιστες πηγές. Οι ασθενείς πρέπει να προστατεύονται και οι πληροφορίες δεν πρέπει υπό καμία προϋπόθεση να διανέμονται απευθείας από τους παρασκευαστές. Επίσης θα πρέπει να, οι πληροφορίες αυτές να καλύπτουν μια δεξαμενή στοιχείων, μια δεξαμενή πληροφοριών. Πιστεύω επίσης ότι δεν θα πρέπει η ενημέρωση αυτή να παρέχεται από τα μέσα ενημέρωσης και πιστεύω ότι πρέπει να ε, αποκλειστούν τα μέσα ενημέρωσης ως παροχής πληροφοριών διότι μπορούν να εκμεταλλευτούν τη θέση τους και την ισχύ τους επιμένω ότι δεν υπάρχει λόγος να παρουσιάσουμε ιδιαίτερα προσκόμματα στο φαρμακευτικό τομέα ούτε χρειάζεται εφόσον παρέχεται ενημέρωση από ιστοσελίδες να γίνει επανέγκριση των ιστοσελίδων αυτών μετά από την υιοθέτηση της, την τροποποίηση της οδηγίας. Ταυτόχρονα πρέπει να εξασφαλίσουμε τον αναγκαίο μηχανισμό ε, για, την, ε, για τους παρασκευαστές ώστε να επιβληθούν κυρώσεις όταν δεν σέβονται τους κανονισμούς. Η EMEA, η ΕΜΕΑ, e e θα πρέπει να είναι ένας από τους ε, φορείς αξιόπιστων, αξιόπιστης μελέτης των ε, προτάσεων και δεδομένου αυτή η οδηγία έχει στόχο, αντολίζεται προς τους καταναλωτές, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις απόψεις των καταναλωτών για να μας εξηγήσουν ακριβώς τι ανάγκες υπάρχουν. Αυτά είναι τα σημαντικά σημεία και τα πιο σημαντικά που ήθελα να σας παρουσιάσω. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις για το, την τροποποίηση αυτή της οδηγίας. Έχω τις τροπολογίες και θα ήθελα να ακούσω σχόλια και παρατηρήσεις. Έχω ανοιχτή προσέγγιση αν υπάρχει οτιδήποτε το οποίο μπορεί να βελτιώσει την πρόταση για να καταλήξουμε σε μια αξιόπιστη, εμπεριστατωμένη και ε, εφαρμόσιμη οδηγία προς όφελος των καταναλωτών. Σας ευχαριστώ κύριε Μπουζόη και τον κύριο Ντεκάμπος. Επίσης ευχαριστώ για τις ε, ε, θαυμάσιες ε, τους εισηγήσεις στις δύο αυτές προτάσεις. Τώρα θα πρέπει να προσέξει τα κείμενα αυτά και η Επιτροπή Περιβάλλοντος, διότι είναι μερικά σημεία τα οποία τους ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και αποτελούν τμήμα των εσωτερικών διαβουλεύσεων. Πρέπει λοιπόν να περάσει η άποψή μας. Ας ακούσουμε τώρα από την κυρία Βάισμπεργκερ και τον κύριο Φόξ και όλοι οι την άποψή τους και την κυρία Γκέπχαρντ. Κυρία Βάισμπεργκερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές ε, για τις εισαγωγικές τους παρατηρήσεις. Συνεργαστήκαμε σαυμάσια και μου αρέσουν. Είμαι πολύ ικανοποιημένη από αυτή τη διαδικασία, δεδομένου ότι όλοι μαζί συνεργαζόμαστε στο θέμα της ενημέρωσης των ασθενών. Πιστεύω ότι εδώ υπάρχει τεράστια ανάγκη ε, να δραστηριοποιηθούμε να κάνουμε κάτι ώστε η ενημέρωση και γραπτή αλλά και προφορική Υπάρχουν πληθώρα πληροφοριών στο διαδίκτυο, οι περισσότερες από αυτές ούτε ελέγχονται, ούτε είναι και καλές, ε, σωστές. Πολλές φορές το, οι και το υγειονομικό προσωπικό αναγκάζεται να διαθέσει 15 λεπτά για να εξηγήσει στον ασθενή ότι όλες αυτές οι πληροφορίες που έχει πάρει από το διαδίκτυο είναι εσφαλμένες και να ξαναρχίσει από την αρχή την όλη εξέταση και την όλη διαδικασία. Υπάρχει λοιπόν μεγάλος κίνδυνος στρέβλωσης των πληροφοριών και της ενημέρωσης. Στην αρχή, όταν ακούστηκαν οι δύο αυτές προτάσεις, υπήρχαν θεμελιώδεις αντιρρήσεις ακόμα και από τις οργανώσεις των καταναλωτών. Όμως, ε, διοργανώσαμε ένα πρωινό εργασίας με εκπροσώπους των διαφόρων ενώσεων και οργανώσεων και ασθενών και καταναλωτών και οι οργανώσεις ασθενών μας είπαν ότι η πρόταση της Κομισιόν ως έχει αυτή τη στιγμή δεν είναι καλή, δεν είναι ικανοποιητική, αλλά πιστεύουν ότι μπορεί να βελτιωθεί και εκεί ακριβώς πρέπει να παρέμβουμε. Εχτες με ξάφνιασε η συζήτηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος διότι από τους σοσιαλιστές και τους πράσινους ακούστηκαν πάρα πολύ σοβαρές επιφυλάξεις και ελέγχθη από τον κύριο Ντάλι ότι θα κάνει μια νέα πρόταση. Να δούμε, να περιμένουμε αν θα τη δούμε. Όμως εμείς αυτή τη στιγμή πρέπει εδώ να διαχειριστούμε τις υπάρχουσες προτάσεις και ο κύριος Ντάλι ίσως ε, μπορέσει να βελτιώσει το κείμενό του, να μην κάνουμε ένα βήμα μπρος και δύο βήματα πίσω. Εγώ πιστεύω αυτά τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή στο τραπέζι μας είναι εξαιρετικά καλά και καλύπτουν πάρα πολλά σημεία, τα οποία αφορούν την ενημέρωση των ασθενών. Όπως είπε και ο κύριος Μπουζόη, βεβαίως διαφημίσεις. Είμαστε εναντίον της ε, διαφημιστικής ενημέρωσης. Πρέπει να υπάρχει σαφή διαχωρισμός μεταξύ πληροφοριών push and pull. Επίσης, ε, όπως είπε ο κύριος Μπουζόη, οι πληροφορίες θα πρέπει να ε, συγκεράσουν μία δεξαμενή πληροφοριών ηλεκτρονικών, μέσω διαδικτύου, μέσω φυλαδίων, μέσω ενημερωτικών δελτίων μέσα στα κουτιά των φαρμάκων. Ο, η ενημέρωση πρέπει να καλύπτει πολλαπλές πηγές. Um, Im Vorfeld eine um, ja wirklich ähm, θα πρέπει επίσης ε, να υπάρχει μία προηγούμενη εξέταση της ενημέρωσης από την EMEA, e e την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να διασφαλιστεί αξιοπιστία. Η εστίαση δεν πρέπει να είναι στην πλευρά του παρασκευαστικού τομέα, αλλά πρέπει να είναι στο πλευρό του καταναλωτή. Εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε, στον καταναλωτή. Έχω και μία ιδέα καινούργια την οποία θα ήθελα να συζητήσω μαζί σας κύριε Μπουζόη. Όσον αφορά το διαδίκτυο υπάρχουν, υπάρχει ενημέρωση σε δύο γλώσσες. Αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπεται στο διαδίκτυο να δημοσιευθεί το χαρτί της, ε, των πληροφοριών που βρίσκεται μέσα ε, στο κουτί των φαρμάκων. Αυτή τη στιγμή αν χάσεις το χαρτάκι αυτό, το διπλωμένο, δεν μπορείς ούτε στο διαδίκτυο να το βρεις, ούτε να σου το στείλει η φαρμακευτική εταιρεία ξανά, οπότε χάνεις τις πληροφορίες. Στην ε, Σουηδία όμως υπάρχει ένα άλλο σύστημα όπου μπορεί κανείς να πληροφορηθεί και για τα φάρμακα αλλά και για τις ε, ασθένειες. Παραδείγματο χάρη, ε, αν πάω στο γιατρό μου ότι έχω ψηλή πίεση, μπορώ να καταφύγω στο διαδίκτυο και να πάρω αξιόπιστες πληροφορίες. Πρέπει λοιπόν να, να υπάρχει μια πλατφόρμα πληροφοριών η οποία να έχει ελεγχθεί και αξιολογηθεί εκ των προτέρων ώστε να μπορώ να πάρω πληροφορίες για τη βασική θεραπεία της, ε, της, της ψηλής πίεσης, παραδείγματος χάρη τους β' αναστολής, τι φάρμακα μπορώ να πάρω, ε, πώς ενεργούν τα φάρμακα, ε, αλλά και επίσης πληροφορίες διατροφής, υγιεινής ζωής, άσκησης κλπ. Πιστεύω λοιπόν ότι ανεξάρτητα από αυτά τα οποία επισημεί ο παρασκευαστικό τομέα, να υπάρχει μια αξιόπιστη, ενημερωμένη και επίκαιρη πλατφόρμα στο διαδίκτυο, από την οποία ο καταναλωτή να μπορεί να τραβήξει, του pool δηλαδή, να τραβήξει, να εξάγει τι ε, πληροφορίε που θέλει. Χωρίς αυτό να αποτελεί βεβαίως διαφήμιση. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, ε, το χρονοδιάγραμμα είμαι ικανοποιημένη. Θα παρακαλούσα όμως να αναβάλουμε λίγο την προθεσμία τροπολογιών, διότι θα ήθελα να διαβουλευθώ και με την Επιτροπή ε, περιβάλλοντος. Πιστεύω ότι εμείς θα πρέπει να είμαστε η δεσπόζουσα επιτροπή εδώ και να λάβουμε τον ηγετικό ρόλο και γι' αυτό θα παρακαλούσα να αναβάλουμε λίγο την ε, τροπολογία, την προθεσμία. Ευχαριστώ πολύ. Θα δούμε τι γίνεται με την πρόθεσμια για τις ε, τροπολογία ε, Αφού ακούσουμε τους κοιόδης ηγητές, έχω μια πρόταση να σας κάνω. Ο κύριος Φόξ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτή την νομοθεσία και να ευχαριστήσω και την κυρία Βάσης Γκέρμπερ και τους δύο εισηγητές για το θέματα. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ του τρόπου με τον οποίο παρέχονται πληροφορίες ε, για τα φάρμακα στους ε, ασθενείς ε, στα κράτη-μέλη. Οι ασθενείς θα πρέπει να, έχουν, να λαμβάνουν ανεωμερωμένε αποφάσεις για τα φάρμακα που τους παρέχονται. Δεν είναι ακριβώς ε, αυτό που λέει η κυρία Βάις Γκέρμπερ ας πούμε. Στη Γερμανία αν χάσετε το ε, φυλάδιο με τις ε, ιατρικές ενδείξεις που περιέχονται στο κουτί δεν μπορείτε το να τα βρείτε στο διαδίκτυο. Συμφωνώ με τους ε, εισηγητές ότι οι πληροφορίες προς τους ασθενείς θα πρέπει να είναι μη διαφημιστικού χαρακτήρα αυστηρός και θα πρέπει να δίνονται μόνο ανεξάρτητες πληροφορίες. Δεν θέλουμε να τους παραπληροφορούμε και δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να δω μια κατάσταση σαν αυτή που έχουμε στι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουμε διαφημίσει την τηλεόραση για φαρμακευτικά προϊόντα. Να σταθώ σε δύο τομείς που με ανησυχούν. Η τροπολογία υπαριθμών 3 για τον κανονισμό, καταρχάς, όλοι γνωρίζουμε εδώ στην Επιτροπή μας ε, τις πιέσεις ε, στον προϋπολογισμό που αντιμετωπίζουν όλα τα κράτη-μέλη και δεν πιστεύω ότι ο φορολογούμενος θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα για αυτό το νέο σύστημα. Ε, είμαι διατεθειμένος να συζητήσω οποιαδήποτε συμβιβασμό για το θέμα, διότι ο οργανισμός θα πρέπει να χρηματοδοτείται καταλήλως, αλλά η άποψή μου είναι ότι η χρηματοδότηση θα πρέπει να προκύπτει από τον κλάδο και όχι από τον φορολογούμενο πολίτη. Με ανησυχεί επίση η τροπολογία 2 και η προσέγγιση που προτείνεται για την ε, ε, πληροφόρηση. Η προσέγγιση αυτή είναι μία για όλους και δεν είναι αναλογική. Είναι άκρος γραφειοκρατική και δεν υποστηρίζω να υπάρχει ρόλος για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για τα προϊόντα αυτά. Να ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε και να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά στα, ε, τους εισηγητές για όσα έκαναν. Η κυρία Ρούλε, παρακαλώ. Ευχαριστώ και τους δύο συγητές εξαιρετικές προτάσεις. Θα πρέπει βεβαίως να συζητήσω με τη συνάδελφό μου αυτή τη στιγμή πάρα πολλές πληροφορίες υπάρχουν στο διαδίκτυο που δείχνει ότι οι καταναλωτές έχουν αυτήν την ανάγκη. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι πληροφορίες είναι και καλές και αξιόπιστες και ελεγμένες, είναι ανεξέλεγκτες. Επίσης, τι πληροφορίες μέσα στο κουτί, στο κουτάκι των φαρμάκων, αν κάποιο χάσει το χαρτάκι αυτό, η μητέρα μου ας πούμε το χάσει ε, και εγώ θέλω να, να ελέγξω, τι είναι αυτό το φάρμακο, τα συστατικά, δοσολογία κλπ. Ε, δεν μπορώ να το, να το λάβω από πουθενά. Ε, είναι εξαιρετικά δύσκολο κάπως ε, να το πάρω πάλι, να μου το στείλουν, να το βρω κάπου. Λοιπόν, αυτό είναι μία δυσκολία μεγάλη. Επίσης, ο διαχωρισμός μεταξύ ε, pull and push και δηλαδή η αποφυγή της ε, διαφήμισης αλλά η παροχή σωστών πληροφοριών είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Καταλαβαίνω βεβαίως ε, την άποψη του κυρίου Φούξ ότι υπάρχει οικονομική στενότητα αλλά ε, στον παρασκευαστικό τομέα και στη φαρμακευτική βιομηχανία υπάρχουν τεράστια περιθώρια ε, χρηματοδότησης αν και εδώ επισέρχεται το θέμα της ουδετερότητος και της των φαρμακευτικών εταιριών. Απ' τη μία έχουν λεφτά, απ' την άλλη όμως δεν είναι και ουδέτερες. Ευχαριστώ. Μιλώ εκ μέρους της συναδέλφου μου, κυρία Μπάρμπαρα, κυρίας Μπάρμπαρα Βάλερ, η οποία είναι σκιώδης, εισηγήτη, αλλά δεν μπορεί να είναι παρούσα εδώ. Οι δύο εκθέσεις αυτές πράγματι είναι πάρα πολύ καλές και εγώ συμφωνώ και Κακολουθούν ένα σωστό ε, διάβλο διότι ζητούν την παροχή πληροφοριών αλλά την παροχή ελεγμένων, αξιολογημένων και αξιόπιστων πληροφοριών προς τον καταναλωτή. Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Επίσης, συμφωνώ με την κυρία Βάις Γκέρμπερ και την κυρία Ρούλη ότι στο ίντερνετ υπάρχει πληθώρα πληροφοριών Και όταν κανείς ε, θέλει να ψάξει για κάτι στο ίντερνετ, ε, ε, βλέπει πάρα πολλές ε, ε, πληροφορίες, ε, διάφορες ιστοσελίδες ενημερωτικές υποτίθεται, αλλά αυτές δεν έχουν ελεγχθεί από κανέναν αξιόπιστο φορέα. Αυτό εμεί που θέλουμε να εξασφαλίσουμε είναι ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες τουλάχιστον είναι ελεγμένες από έναν φορέα, από ουδέτερο και αξιόπιστο ώστε να μην στρεβλώνουν τις απόψεις του καναλωτού και στο τέλος της γραφής μπορεί να είναι και επικίνδυνες. Συμφωνώ με την κυρία Ρουλή ότι θα πρέπει να φροντίσουμε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων να είναι ανεξάρτητος και να μην επηρεάζεται από την παρασκευαστική βιομηχανία, από τις φαρμακευτικές εταιρείες, πρέπει να είναι ουδέτερη, να τηρεί μια ουδέτερη στάση. Ελπίζω να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και την ε, ποιότητα των εργασιών αυτού του οργανισμού, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, ο οποίος ε, μέχρι τώρα λειτουργεί αλλά δεν μας έχει και ενθουσιάσει. Ελπίζω στο μέλλον να ανεβεί η ποιότητα των εργασιών του. Όσον αφορά τώρα την έξεση, την πρόταση του κυρίου Μπουρζόη, η κυρία Βάιλερ συμφωνεί με τον προσανατολισμό του, πιστεύει ότι οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση και υποστηρίζουμε τις ε, προτάσεις σας. Πιστεύω ότι στις τροπολογίες σας θα υπάρχει ένα θετικό σήμα, δηλαδή θα υπερψηφιστούν, δεν νομίζω να υπάρχει ένα πρόβλημα με τις τροπολογίες σας. Ένα πράγμα μόνο έχω να παρατηρήσω, ότι η οδηγία αυτή ισχύει μόνο για φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κρίμα που δεν καλύπτει όλα τα φάρμακα με η άνευ ιατρική συνταγής. Επίσης χρειαζόμαστε μία, ένα σαφή ορισμό των ψευδεπίγραφων φαρμάκων και μία εκστρατεία ενημέρωσης για τους καταναλωτές για να ξέρουν ακριβώς ποιες είναι οι πηγές σωστής πληροφόρησης και, για το, και επίσης για να τους επιστήσουμε την προσοχή στον κίνδυνο ε, των ε, ψεύτικων, των ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών. Αυτές τις παρατηρήσεις ε, είχα να πω εκ μέρους του συναδέλφου μου και του συγχαίρω για την εξαιρετική εργασία και τους δύο συγητές. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Μόνο μία παρατήρηση για τις πληροφορίες στο διαδίκτυο για τα φάρμακα. Να σας υπενθυμίσω ότι στην έκθεσή μου για τις καθολικές υπηρεσίες, τα δικαιώματα και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες οι ρυθμιστέ τηλεπικοινωνιών των κρατών μελών μπορούν να απαιτήσουν να διαβιβάζονται μηνύματα δημοσίων υπηρεσιών και νομίζω ότι τα φαρμακευτικά θέματα είναι τομεί ε, μέσω των, οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη διο, το διάβλο επικοινωνία. Αν για παράδειγμα όλα τα κράτη, οι μέλη θέλουν να ενημερώσουν τους χρήστες του διαδικτύου για τα ε, πιστοποιημένες ιστοσελίδες τις οποίες θα μπορούσαν να βρουν πληροφορίες. Αν θέλει, δεν ξέρω, οι συγητές να τα αναφέρουν, θα μπορούσα να τους δώσω περαιτέρω λεπτομέρειες. Έχουμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ, ο οποίος παρακολουθεί το θέμα στενά. Προτείνω να του δώσουμε το, λίγο, το λόγο να μας πει τι έχει να μας πει και μετά θα ζητήσω από τον ε, καθηγητή Ντεκάμπος και από τον κύριο Μπουσόη να συνοψίσουν τη συζήτησή τους και ε, να συμφωνήσουμε λίγα πράγματα και για το χρονοδιάγραμμα. Παρακαλώ, εκπρόσωπος της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συζητητές για την πολύ καλή συνεργασία και τα θετικά σχόλια τα οποία μας ενθαρρύνουν, τα οποία είναι σερεντικά για, την Κομισιόν. Ιδίω ε, σε ό,τι αφορά τις ε, βασικές αρχές στις οποίες πρέπει να στηρίζεται η, οδηγία αξιοπιστία, κατανόηση να είναι κατανοητή, ε, ουδέτερη, η αρχή της ουδετερότητας, Ο νέος μας Επίτροπος δήλωσε κατά την ακρόαση του στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ότι θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή ε, στην, στον καταναλωτή. Οι νέες προτάσεις θα ε, εστιάζονται, θα απευθύνονται δηλαδή ε, στον καταναλωτή και οι προτάσεις αυτές δεν αντιπροσωπεύουν μία επιστοδρόμηση ίσα ίσα επιδιώκουν να βελτιώσουν και να διευρύνουν την νομοθετική διαδικασία. Ελπίζω να μην υπάρχει καμία παρανόηση όσον αφορά αυτές τις δηλώσεις του Επιτρόπου. Ο κύριος ε, <clears throat> Ντάλι, ο Επίτροπος, ο αρμόδιος ε, Επίτροπος ε, πιστεύει και έδωσε τις διαβεβαιώσεις του ότι θα ενισχύσει τα θέματα της προστασίας, αξιοπιστίας και ουδετερότητας δεν πιστεύω να υπάρχει καμία παρεξήγηση και να ερμηνεύτηκαν οι δηλώσεις του ως επιστοδρόμηση. Ίσα ίσα δεσμεύτηκε να ενισχύσει τη διάσταση των καταναλωτών. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να εκφράσουμε τη θέση μας ε, με μονομένων θεμάτων, όμως Βλέπω στη συζήτηση και σημείωσα πολλές ιδέες που πρέπει να συζητηθούν. Παραδείγματο χάρη η διασύνδεση με την, την υπάρχουσα τράπεζα δεδομένων και την ιδέα της κυρίας Βάισμπεργκερ εάν μέσω πυλών του διαδικτύου μπορέσουμε για τους ασθενείς και τους καταναλωτές να παράσχουμε καλύτερες και πιο εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες μέσω μιας πλατφόρμας ε, συγκεντρωτικής και περιεκτικής αντί της πληθώρας των ιστοσελίδων από διάφορες ανεξέλεγκτες πηγές. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να εκφράσω την απόψή μου, όμως σημείωσα αυτές τις απόψεις, αυτές τις παρατηρήσεις. Το... Η Επιτροπή σας, η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς, ε, πάντοτε λαμβάνει υπόψη και εξετάζει εις βάθος τις ε, προτάσεις μας και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μια οδηγία η οποία θα ρυθμίζει επιτυχώς το θέμα της ενημέρωσης των καταναλωτών. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Να ζητήσω τώρα από τους δύο συγχυτές να συνοψίσουν και να πω πρώτα κάτι για το χρονοδιάγραμμα να σας κάνω μια πρόταση και μετά να το σχολιάσετε. Προτάθηκε να χρησιμοποιήσουμε λίγο παραπάνω χρόνο για τις τροπολογίες και να δώσουμε και στους ηγητές λίγο περισσότερο χρόνο να συνεργαστούν με τους κοιόδης ηγητές διότι οι πληροφορίες που έχουμε εμείς ε, και νομίζω ότι θα σας επιβεβαιώσετε κι εσείς ε, ότι είναι ότι η ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος θα γίνει τον Ιούνιο και επομένω ε, αυτό θα συζητηθεί μάλλον στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Επομένω, μπορούμε να προτείνουμε να έχουμε προθεσμία για τις τροπολογίες 31 Μαρτίου και κατόπιν να εξετάσουμε τις τροπολογίες στι 27 Απριλίου και ψηφοφορία στι 28 Απριλίου. Αυτό στη συνέχεια θα σας δώσει ένα μήνα για να διαπραγματευτείτε με την Επιτροπή περιβάλλοντο ώστε να περάσει και η θέση μα. Αυτή είναι η πρόταση. Να ζητήσω λοιπόν και από του δύο εισηγητές, οι συντάκτε, ε, αν θέλετε τεχνικώ, είστε συντάχνε. να μα πείτε αν συμφωνείτε και με αυτή την πρόταση για το χρονοδιάγραμμα. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Κορέια Ντεκάμπο και στη συνέχεια θα πάρει το λόγο ο κύριος Πουσόη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με το χρονοδιάγραμμα. Αν ε, διευρύνεται και η προθεσμία είναι ακόμα καλύτερα για μας. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσον αυτός ο περισσότερος χρόνος θα μας ε, βοηθήσει να επιλύσουμε τις διαφορές μας. Αλλά τέλος πάντων ε, όσο περισσότερος χρόνος τόσο το καλύτερο. Από τα όσα ακούσαμε στη συζήτηση παρά το γεγονός ότι εγώ ήμουν αυτός ο οποίος είπα ότι τα θέματα αυτά είναι λίγο απλά, είναι σχετικά σύντομα, ε, σας εξέφρασα μόνο την άποψή μου για τη δική μου τη γνωμοδότηση. Είμαι όμως και σκιώδης γιατί για τη ε, γνωμοδότηση του κυρίου Μπουσόη και δεν εκφράστηκα γι' αυτό και φαντάζομαι ότι το ίδιο έκανε και ο κύριος Μπουσόη. Ε, επιτρέψτε μου λίγο να κάνω κάποια σχόλια λοιπόν για την οδηγία. Πρώτον, συνεργαστήκαμε και κάποιες από τις ε, προτάσεις μου έχουν ήδη συμπεριληφθεί στο κείμενο του κυρίου Μπουσόη, τον οποίο και ευχαριστώ γι' αυτό. Θεωρώ ότι αυτό είναι και απόδειξη καλού συντονισμού. Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία όμως θα πρέπει ίσως να διευκρινίσουμε περαιτέρω. Το πιο σημαντικό είναι η δυνατότητα που δίνεται από την οδηγία στον φαρμακευτικό τομέα να ενημερώνει περαιτέρω τους ε, καταναλωτές. Αλλά αυτό ουσιαστικά αποδεσμεύει τον φαρμακευτικό τομέα από την ευθύνη που έχουν για τις πληροφορίες που δίνουν. Και αυτό κατεμένα παράδεκτο. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε φορείς οι οποίοι θα εξειδικεύονται στο έργο τους. Και φυσικά Φαντάζομαι ότι ο κλάδος δεν ενδιαφέρεται και ιδιαίτερα ο κάθε παραγωγός ε, να ε, κάνει αυτή τη δουλειά γιατί αυτό θα έχει επιπλέον άχθος. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι μπορούν να το ξεφορτωθούν αυτοί και να το φορτώσουν κάπου αλλού. Θα πρέπει ο κλάδος να αναλάβει και τις ευθύνες του και αν ε, ε οι αρμοδιότητες αλλού ε, δεν θα έχουν και καμία ευθύνη. Δεν λέμε ότι ο φαρμακευτικός κλάδος ε, δεν έχει ποτέ ευθύνη, αλλά είχαμε και κάποια πρόσφατα περιστατικά με αντικαταθλιπτικά, για παράδειγμα, στα οποία είχαμε πολύ σοβαρές περιπτώσεις και θανάτους ακόμα και αυτό δεν μπορούμε να το αφήσουμε να περάσει έτσι. Δεν μπορεί ο φαρμακευτικός κλάδος να μην έχει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που δίνονται γιατί θα έχει εκχωρήσει αυτή την αρμοδιότητα σε κάποιο τρίτο. Είμαστε λοιπόν κατά αυτής της δυνατότητας. Εάν, ε, για παράδειγμα, ε, δεν υπάρχει υποχρέωση του ιατρού να ενημερώνει τον ασθενή, τα πράγματα πηγαίνουν ακόμα περισσότερο. Δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε το δικαίωμα στον ιατρό να κάνει μια προσωπική συζήτηση όπως γίνεται συνήθως από τον καιρό του Ιπποκράτη, άλλωστε με τον ασθενή του. Για τις προφορικές ε, απαντήσεις. Ο εισηγητής λέει ότι η δυνατότητα αυτή θα μπορεί να αντικαταστήσει την γραπτή ενημέρωση. Για παράδειγμα, ότι θα μπορούν να δοθούν προφορικές ε, πληροφορίες από τηλεφώνου. Το να λέμε ότι μπορούμε να δούμε πληροφορίες παντού είναι σαν να περνάμε από το 0 στο 100. Ε, ξαφνικά. Ε, εάν για παράδειγμα στη Γερμανία δεν μπορεί κάποιο να βρει τις πληροφορίες στο διαδίκτυο, τώρα αυτή τη στιγμή θα μπορεί να τις πάρει από το τηλέφωνο, αλλά ποιο θα μας εγγυάται ότι είναι σωστέ αυτές τις πληροφορίες. ελοχεύει φυσικά ο κίνδυνος αυτές οι ε, πληροφορίες να γίνουν πληροφορίες ε, τύπου διαφήμισης. Και φυσικά εδώ ε, διστάζουμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Όσον αφορά τώρα τα σχόλια τα οποία έγιναν. σε γενικές ε, γραμμές ε, συμφωνούμε νομίζω όλοι να ευχαριστήσω όλους όσους παρενέβησαν να κάνω όμως μια ερώτηση προς την Κομισιόν ε, δεδομένου ότι είναι παρούσα εδώ όσον αφορά σε αυτό το θέμα της ε, αυτορύθμισης και της ρύθμισης. Στην ε, Σουηδία υπάρχει, ένα, ε, υπάρχει δυνατότητα αυτορύθμισης, αλλά... Υπάρχει και δυνατότητα παρέμβασης από πλευράς δημοσίου. Υπάρχει μια κοινοπραξία ιδιωτικού, δημοσίου και ιδιωτικών φορέων και επομένως αυτή δεν είναι αυτορύθμιση αυτή καθεαυτή, είναι συρρύθμιση. Επομένως, στο κείμενο της ε, Κομισιόν αυτό θεωρείται αυτορυθμιστικό αλλά δεν είναι. Και υπάρχει και μια αμφισημία σημειολογική η οποία μου φαίνεται προβληματική και επομένως ζητώ διευκρινήσεις. Ελπίζω, λέει ο Πρόεδρος, να έχουμε χρόνο. Ε, διαφορετικά θα το κάνουμε μετά. Ο Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, και για τα θετικά σχόλια και για την επικοδομητική ε, ε, προσέγγιση. Εργάστηκα στενά με τον κύριο Κάμπος και τον ευχαριστώ πολύ για τα όσα είπε βεβαίως θα λάβω υπόψη μου τις παρατηρήσεις του και τα σχόλιά του σχετικά με την διατηλεφώνου, με την λεκτική δηλαδή συλλογή ε, πληροφοριών. Ε, όταν έρθει η στιγμή θα το ε, λάβω υπόψη μου. Νομίζω αγαπητοί συνάδελφοι ότι πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι θέλουμε να καταργηθεί πλήρως η διαφήμιση ε, για τα φάρμακα και επίσης θα πρέπει να κάνουμε και μια σαφέστατη, ε, έναν σαφέστατο διαχωρισμό ανάμεσα στις πληροφορίες τύπου pull και τύπου push. Επίσης ε, να εμπλέξουμε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, δηλαδή να ελέγχουν τις κρυφές διαφημίσεις ε, έτσι ώστε να τα χρησιμοποιήσουμε με δύο τρόπους, δηλαδή και για να προωθήσουμε ε, τη σωστή ενημέρωση και για να καταργήσουμε την κρυφή διαφήμιση. Uh, free information for uh, are allowed in uh, ε, ε, σχετικά με τα φάρμακα χωρίς ε, συνταγή, ναι, στη χώρα μου πρέπει να πω ότι επιτρέπεται η διαφήμιση για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα και νομίζω ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν κάποια στιγμή και αυτά στην οδηγία. Το θέμα των φαρμάκων ε, ε, πρέπει να αποτελεί βεβαίως ε, και ένα θέμα σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στον ασθενή και τον γιατρό Γι' αυτό λοιπόν πιστεύουμε ότι από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσουμε ε, και εν πάση περιπτώσει η πληροφόρηση που θα δίνεται θα πρέπει να είναι ουδέτερη πληροφόρηση για τα διάφορα φάρμακα και οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να ακολουθούν και, τον, ε, το φάρμακο. Τώρα, επιπλέον πληροφορίες όντως μπορούν να βρεθούν και στο διαδίκτυο κτλ και κατά τα λοιπά συμφωνώ με τον κύριο Δεκάμπος όχι μόνο γιατί έχω σπουδάσει ιατρική αλλά γιατί πραγματικά πιστεύω ότι είναι εμβληματική, είναι ουσιώδης η σχέση ανάμεσα στο γιατρό και τον ασθενή και θα πρέπει να παραμείνει. Ευχαριστώ την κυρία Γκέμπχαρντ η οποία αν κατάλαβα καλά μου υποσχέθηκε ότι θα περάσουν ε, οι περισσότερες τροπολογίες από την ομάδα της οποίας ηγείται εδώ στην Επιτροπή μας. Όσον αφορά τώρα την υποχρέωση των προμηθευτών για δημόσια πληροφόρηση, ε, θα σκεφτώ και θα ε, δω το κείμενο το οποίο θα μπορούσαμε να υποβάλουμε ως τροπολογία. Τέλος, συμφωνώ απολύτως με το νέο χρονοδιάγραμμα πιστεύω ότι αυτές οι 12 επιπλέον μέρες θα μας επιτρέψουν να σκεφτούμε καλύτερα τις τροπολογίες αλλά και να διαπραγματευτούμε αποτελεσματικότερα και με αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας με την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής ε, ε, θα ε, να μας απαντήσει παρακαλώ στη συγκεκριμένη ερώτηση, στη που έθεσε ο καθηγητής Δεκάμπος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η πρόταση οδηγίας μας προβλέπει ότι καταρχήν θα πρέπει να υπάρξει επίσημος έλεγχος των πληροφοριών που διαχέονται αλλά υπάρχει και μια παράγραφος η οποία αφήνει και ένα περιθώριο ελιγμών και πράξεων στα κράτη-μέλη ε, έτσι ώστε να εμπλέξουν αυτορυθμιστικά ε, ή συνρυθμιστικά σώματα. Αυτές ε, είναι οι αρμόδιες ε, ε, αρχές αποτελούν το σκέλος της αυτορύθμισης από όσο κατανοούμε εμείς και η βιομηχανία αποτελεί το σκέλος της συρρύθμισης. Επομένως το κράτος μέλος έχει την δυνατότητα βάσει του περιθωρίου που αφήνει η οδηγία να συζητήσει με τις αρχές αυτορύθμισης ή συρρύθμισης. Επίσης είναι γεγονός ότι το πρότυπο της Σουηδίας είναι συνρυθμιστικό και όχι αυτορυθμιστικό. Έχετε δίκιο. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε εκπρόσωπο της Επιτροπής. Ευχαριστούμε και όλα τα μέλη τα οποία ε, πήραν μέρος στη συζήτηση αυτή. Τώρα θα σταματήσουμε για δύο-τρία λεπτάκια έτσι ώστε να φτάσει ακριβώς 10 και θα αρχίσουμε να ψηφίζουμε. Να σας πω ότι θα έχουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία γιατί έχουμε πολλές ε, τροπολογίες. Γι' αυτό λοιπόν σιγουρευτείτε ότι έχετε έτοιμες τις κάρτες σας, ότι είστε έτοιμο πόλεμοι. Ναι, ναι, ε, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε βλέπω στην βουλγαρική μετάφραση ότι υπάρχει διαφορά στο όνομα της οδηγίας. Ε, συνήθως χρησιμοποιώ το αγγλικό κείμενο, αλλά στο αγγλικό κείμενο γράφει medicinal products κτλ. κτλ ενώ ενώ στα βουλγαρικά λέμε <clears throat> ε, ε, ιατρικά σκευάσματα τα οποία έχουν συνταγογραφηθεί για ανθρώπινη και ζωική χρήση, κάτι τέτοιο είναι ένα μπλεγμένο πράγμα το οποίο εν πάση περιπτώσει δεν μεταφράζει σωστά την, ε, τον τίτλο της οδηγίας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Θα το δούμε, θα, θα, θα κάνουμε την απαραίτητη διόρθωση. Διάλειμμα λοιπόν μέχρι τις 10.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 Right, Καθίστε παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι, θα προτιμούσα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Παρακαλώ, ησυχία. Τι γίνεται τώρα, τα, τα συμφωνείτε για πώς θα ψηφίσετε. Παρακαλώ, ησυχία δεν θα, συμφω... χρησιμοποιήσουμε το ηλεκτρονικό, την κάρτα μας για όλες τις ψηφοφορίες, μόνο εκεί που είναι κλειστή η ψηφοφορία. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν την ηλεκτρονική ψηφοφορία όπου δεν είναι πολύ καθαρό το αποτέλεσμα, ε, για να τσεκάρουμε. Λοιπόν, για τσεκάρετε παρακαλώ τις κάρτες σας και βάλτε την κάρτα σας μέσα στο, στο μηχανάκι. 26 έχουμε, 26 μέλη έχουμε προς το παρόν. Για να τσεκάρουμε σας παρακαλώ το σύστημα. should come up with a, um, Λοιπόν, ο τεχνικός επαναρρυθμίζει το σύστημα. Ένα λεπτό, περιμένετε παρακαλώ, να, φτιαχ... φτιαχτεί η τεχνολογία. Παρακαλώ πολύ, για να τσεκάρουμε τον αριθμό των μελών. Βάλτε... Παρακαλώ, κάντε μια δοκιμαστική ψηφοφορία υπέρ ή κατά, ό,τι θέλετε. Έτσι, τσεκάρουμε απλώς τον αριθμό των παρόντων, των μελών. Άρχεται η ψηφοφορία που λέμε. Πιέστε το κουμπάκι. working here, all right. No. All right. All right, let's clear the and start again then. Να ξαναρχίσουμε, ξανά, ξανά. Εντάξει είναι τώρα δουλεύει. Δεν δουλεύει, δεν δουλεύει το σύστημα λέει ένα μέλος. Γενική... Γενικώ ορισμένα δεν δουλεύουν. Λοιπόν, παρακαλώ όσοι θέλουν να ψηφίσουν, βάλτε την κάρτα σας τώρα, λέει ο πρόεδρος, τώρα. Ωραία. Η μπροστινή σειρά φαίνεται έχει πρόβλημα. Can you, clear, can you close the vote now? Right. Right, look, let's just have one more time. Άλλη μια φορά. Βάλτε παρακαλώ την κάρτα σας όσοι θα ψηφίσετε. Άλλο ε, ένα τσεκάρισμα. Να, δεν δουλεύει. You should have a... Is your card in properly? Right. Είναι σωστά η κάρτα σας μέσα στο σύστημα. Τη βάλατε σωστά. We can only allow a certain amount of time. Άλλη μία, άλλο ένα τσεκάρισμα παρακαλώ. Τελευταίο. Λοιπόν, να, να ελέγξουμε τους αριθμούς. Όλα τα μέλη του ΕΛΚ, παρακαλώ του ΕΛΚ, ψηφίστε τώρα. Υπέρ, λέει ο πρόεδρος. Όλα τα μέλη του ΕΛΚ, του ΕΛΚ και μόνον, ψηφίστε τώρα. Ο κύριο Δε Κάμπο ε, πήγε στο πλευρό των, ε, του ΕΛΚ αυτή τη στιγμή. Μπράβο, μπράβο. So, so, uh, I've closed the vote on the EPP. Λοιπόν, τελειώνουμε με το ΕΛΚ. 12. 13. 13 μέλη του ΕΛΚ, εντάξει. Τώρα να δοκιμάσουμε τους ε, σοσιαλιστές και, ε, και δημοκράτες μόνο παρακαλώ σοσιαλιστές και δημοκράτες αν δεν δουλεύει καθίστε αλλού λέει ο πρόεδρος so, the vote is open for all S&D members S&D λοιπόν and the vote is closed τελείωσε η ψηφοφορία και έχουμε 9, 10, 10 ωραία Τώρα, οι φιλελεύθεροι, παρακαλώ μόνο οι φιλελεύθεροι να ψηφίσουν. Μόνο οι φιλελεύθεροι. Τέλος της ψηφοφορίας. Τέσσερις φιλελεύθεροι, ωραία. Η πράσινη. Όχι, δεν δουλεύει το σύστημα. Εκεί που κάθεστε, πράσινη, ομάδα των πρασίνων. Can you check um, Ελέγξτε παρακαλώ το, την ε, κάρτα, την ηλεκτρονική, το σύστημα. Έλεγα ότι με την ηλεκτρονική ψηφοφορία θα κερδίσουμε χρόνο. Αλλά εδώ έχουμε χάσει πάρα πολύ χρόνο με όλη αυτή την, ε, τα τεχνολογικά προβλήματα. Αντί να κερδίσουμε, χάνουμε χρόνο. Right, so the vote is... Λοιπόν, πράσινη, γκουε και συντηρητική. Πράσινη, γκουε και συντηρητική. Παρακαλώ ελέγξτε το σύστημα, το μηχανάκι, έληξε η ψηφοφορία. Ωραία. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η πρώτη ψηφοφορία αφορά την έκθεση της κυρίας Γκέρμπερ. Πού είναι η συγκήτρια? Ε, θέλετε να πείτε κάτι, καμία παρατήρηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Πρόκειται για την απλούστευση της γραφειοκρατίας, βελτίωση της νομοθεσίας μέσω του κανονισμού. Είναι οχτώ οδηγίες της μετρολογίας, τις οποίες θέλουμε να καταργήσουμε, αλλά δεν θέλουμε να δημιουργηθεί ένα νομικό κενό, απλώς θέλουμε να απλουστεύσουμε τη διαδικασία επειδή υπάρχει γενική οδηγία, έχουμε ε, παρουσιάσει μια πάρα πολύ καλή πρόταση την οποία δέχεται και το Συμβούλιο υπήρχαν διαφορετικές προτάσεις από την κυρία Γκέμπαρτ και από μένα η ιδέα όμως και ο στόχος είναι ο ίδιος απλώς το παρουσιάσαμε διαφορετικά μίλησα με την νομική υπηρεσία μου είπε τη μορφή με την οποία πρέπει να παρουσιάσουμε την πρόταση τελικά επιτύχαμε συμφωνία και μπορούμε ξεκάθαρα να δώσουμε ένα μήνυμα στο Συμβούλιο ότι ε, θα επιτευχθεί, θα, επιτευχθεί μια διαθεσμική συμφωνία. Ε, ευχαριστώ και την, για την υποστήριξη των σκιωδών εισηγητών και είμαι αισιόδοξη ότι θα κάνουμε έναν ε, επιτυχή τρίλογο με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ για την εργασία που έχετε κάνει. Ψηφίζουμε. Α, κυρία Γκέμπαρτ, ευχαριστώ. Ναι, σωστά πηγαίνουμε προς την ίδια κατεύθυνση και προσπαθήσαμε να βρούμε διαφορετικές ε, μεθόδους ε, εφαρμογής. η κατάργηση ή η ελάφρυνση της ε, γραφειοκρατίας είναι ένας επιθυμητός στόχος αλλά είναι δύσκολος να επιτευχθεί δεδομένου ότι εδώ εμπλέκονται στοιχεία αμοιβαία αναγνώρισης και είχαμε μεγάλες δυσκολίες να ε, συμφωνήσουμε στην κατάργηση όλων αυτών των οδηγιών, οχτώ οδηγίες. Γι' αυτό προτείνω να το συνδυάσουμε με την ε, Κομισιόν, αυτό το οποίο έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα παρουσιάσει μια οριζόντια οδηγία. Τώρα, η νομική υπηρεσία λέει αυτό δεν είναι δυνατό να γίνει εγώ όμως ξέρω άλλες πτυχές της νομοθεσίας όπου έχουν καταργηθεί παλαιότερες οδηγίες σε βάση του άρθρου 6 και έχει παρουσιαστεί οριζόντια οδηγία από την Κομισιόν. Τώρα γιατί σε αυτό το θέμα της ε, μετρολογίας δεν είναι δυνατό να γίνει δεν ξέρω. Τώρα, εάν η πρόταση αυτή δεν περάσει, θα πρέπει να ψηφίσουμε την ε, τροπολογία 14. Δεν θα παρουσιάσω προφορική τροπολογία η οποία δεν μας ε, βοηθάει, διότι ξέρω ότι οι περισσότεροι συμφωνούν με τις τροπολογίες. Βεβαίως, επί της ουσίας, συμφωνώ με την πρόταση της κυρίας Βάισμπεργκερ που θέλει να αντικαταστήσει το 2013 με το 2014 και θα ήθελα ε, να γραφτεί στα πρακτικά. Εάν περάσουν οι τροπολογίε της κυρίας Βάισμπεργκερ, τότε θα συμφωνήσουμε επί της εξαίσεως γενικά ή πω τον όρο ότι αυτά τα οποία έχει ανακοινώσει η κυρία Βάισμπεργκερ θα περάσουν μέσω του τριλόγου και θα γίνει μία αναθεώρηση πριν από αυτή την ημερομηνία πριν από αυτή τη χρονολογία, 2012-2013. Για να επιτύχουμε μία συμφωνία των θεσμικών οργάνων. Εάν λοιπόν υπάρξει αυτή η αναθεώρηση και την αποφασίσουμε μέσω του τριλόγου, τότε θα μπορέσουμε να υπερψηφίσουμε την έκθεση. Όμως θα ψηφίσουμε την τροπολογία 15 η οποία είναι από την ομάδα μου και αυτό μου το ζήτησε η ομάδα μου και θα ήθελα παρακαλώ να, την ψηφίσουμε. Την τροπολογία 15. Ευχαριστώ. Η Νομική Επιτροπή είπε ότι δεν μπορούμε να θέσουμε όρους και δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε μία αναθεώρηση η οποία ακόμα δεν υπάρχει. Όμως είναι σωστό. Μέσω της διαθεσμικής ε, συμφωνίας μπορούμε στην αναθεωρημένη οδηγία να γίνει μία παραπομπή και αν με την τροπολογία αυτή πάρουμε μία παράταση α, ενός ακόμα έτους από το 2014 ε, πιστεύω ότι θα επιτύχουμε το στόχο μας και σας ε, υπόσχομαι ότι μέσω του τριλόγου, δηλαδή της ε, διασεσμικής ε, διαβούλευσης, ε, θα περάσει αυτό το θέμα. Ευχαριστώ τους, την συγγήτρια και τους κοιόδης. Και επίσης πριν δώσουμε την τελική μας έγκριση έχουμε συμφωνήσει να ζητήσουμε μία δήλωση από την Κομισιόν. εάν ε, στο θέμα των νομικών ε, προσκομμάτων ε, στα, τα οποία μας είπε το Συμβούλιο, η νομική υπηρεσία. Λοιπόν, ψηφίζουμε την πρώτη τροπολογία 5, Weisberger, δεκτή. Τροπολογία 15 άρθρο 1, ηλεκτρονική παρακαλώ, για την τροπολογία 15 ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τέλος, πέρας της ψηφοφορίας. I απορρίφθηκε, απορρίφθηκε. Ναι, σα, σαφώς. Μία ψήφος υπάρχει 23 κατά. Απορρίφθηκε. Η τροπολογία 15. Προχωρούμε στην τροπολογία 14 Βάσκερμπερ υπέρ κατά ε, δεκτή. Και ε, καταπίπτει η τροπολογία 6, άρθρο 1α νέο, τοπολογία 7 της εισηγήτριας υπέρ κατά δεκτή. Τώρα, αν κατάλαβα σωστά, η κυρία Γκέπαρτ δεν εμένει στην ε, προφορική της τροπολογία, οπότε Προχωρούμε, προχωρούμε έχοντας υιοθετήσει την 14, η 16 και η 8 είναι και, εγκρίνονται και αυτές, δεν ψηφίζονται. Προχωρούμε στη σελίδα 6, 6 ε, τροπολογία 12, κρίσιμη τροπολογία. Έχουμε το εκτιμώντας 6, τροπολογία 12 της κυρίας Γκέπαρτ, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τροπολογία 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, ε, πέρα ψηφοφορίας απερίφθη 10 υπέρ 23 κατά απερίφθη τροπολογία 2 Βάσκερμπερ υπέρ κατά δεκτή 3 Βάσκελμπερ υπέρ α Συγγνώμη λέει ο πρόεδρος. Λάθος. Όλα τα άλλα δεν θα ψηφιστούν. Τελική ψηφοφορία της, του σχέδιου έκθεσης υπέρ. Υπέρ. Κατά. 30 υπέρ. Ε, τρεις αποχές. Συγχαρητήρια κυρία Βάις Γκέρμπερ και σας εύχομαι κάθε επιτυχία και δύναμη στις ε, διαβουλεύσεις σας με το Συμβούλιο. Προχωρούμε τώρα στην γραμμολόγηση για τα διανοητικά δικαιώματα. Η κυρία Ρόιτοβα. Θέλετε να σχολιάσετε μήπως τίποτα πριν αρχίσει η ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω όλους ε, όσους συνεργάστηκαν μαζί μου σε αυτό το περίπλοκο θέμα. Θα πρέπει να παλέψουμε για την έκθεση αυτή στην Επιτροπή Νομιθωκών Υποθέσεων. Έχουμε πάρα πολλές τροπολογίες και έχει αναβληθεί η ψηφοφορία για ένα μήνα. Όμως, θα πρέπει και εδώ να αποφασίσουμε ε, πού μπορούμε να ζητήσουμε κατά τμήματα ψηφοφορία και πού δεν μπορούμε. Διότι σε κάποιες ε, περιπτώσεις ε, ακούστηκε ότι δεν μπορούμε να ζητήσουμε κατά τμήματα ψηφοφορίας εγώ όμως θα ήθελα να έχουμε ε, κατά ψηφοφορίας ε, σε μια τροπολογία που πρότειναν οι σοσιαλιστέ και οι δημοκράτες. Επίσης υπάρχει ένα λάθος ε, στο κατάλογο ψηφοφοριών για τις τροπολογίε 30 και 31. Κάποιοι έχετε συν και κάποιοι έχετε πλην. Ε, αλλά και η συγγήτρια και το ΕΛΚ υποστηρίζουν αυτέ τι τροπολογίε. Διότι η συμβιβαστική πρόταση η οποία η υπήρξε αντικείμενο συμφωνίας ε, αποσύρθηκε. Δεν θέλω να καθυστερήσω άλλο γιατί είναι περίπλοκη αυτή η ψηφοφορία, επομένως αφήνω να ψηφίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Από ό,τι βλέπω υπάρχουν αρκετές συμβιβαστικέ τροπολογίες οι οποίες κατατέθησαν και θα τις προσέξουμε κατά την ψηφοφορία. Θα ήθελα να ενημερώσω όλους ότι καταρχάς ε, η συνεδρίαση αυτή μεταδίδεται στο διαδίκτυο αλλά έχουμε και ένα τηλεοπτικό συνεργείο από το κανάλι του Κοινοβουλίου που κάνει ένα ρεπορτάζ για τις συνεδριάσεις. Γι' αυτό λοιπόν προσέχουν πάρα πολύ τη δουλειά της Επιτροπής μας. Ε, θα έπρεπε να χαιρόμαστε. Είναι παρόντες εδώ στην αίθουσα, τους βλέπετε άλλωστε. Κυρία Ράπτη, θέλετε το λόγο. Κυρία Ράπτη, θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ήθελα πριν προχωρήσουμε στην ψηφοφορία να ευχαριστήσω την κυρία Ρόιτοβα και τους υπολείπους συναδέλφους για τη συνεργασία που είχαμε. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική γνωμοδότηση που θα βοηθήσει πάρα πολύ το ευρωπαϊκό τοπίο. Ε, θέλω να επιστήσω την προσοχή στα εξή. Πρώτον, θεωρώ θετικό πρέσαμε να κάνουμε κάποιες, να καταλήξουμε σε κάποιους συμβιβασμούς. Δεν ήταν εύκολο και έχουν και πολλά ακόμα να γίνουν. Ε, θέλω να επισημάνω επίσης ε, μερικά πράγματα, αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, να υπογραμμίσω ότι έχουμε καταλήξει στην ανάγκη ελέγχου της αποδοτικότητας της νομοθεσίας που ισχύει και των παραβιάσεών της και προσανατολιζόμαστε στο αίτημα για να θεσπιστούν επιπλέον μέτρα μέχρι, να φτάνουν μέχρι και ποινικέ κυρώσεις στην περίπτωση που διακυδεύονται ανθρώπινες ζωές. Να υπογραμμίσω όμως ότι το αίτημα αυτό συνοδεύεται πάντα και σε σημεία στα περισσότερα σημεία του κειμένου από την απέτηση να γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα κυρίως της ιδιωτικότητας. Αισθάνομαι την ανάγκη να το τονίσω αυτό ιδιαίτερα γιατί γνωρίζω ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την προηγούμενη περίοδο έχει ε, δοθεί μάχη. Ε, μάχη στην οποία μάχη πρωταγωνιστές ήταν άνθρωποι που βρίσκονται και μέσα σε αυτή την Επιτροπή σήμερα. Πολύ σημαντική θεωρώ επίσης τη νέα παράγραφο που προτείνεται για την ευαισθητοποίηση του κοινού. Και αυτό γιατί μόνον ο ενημερωμένος καταναλωτής είναι σωστός καταναλωτής. Ε, έχω κάποιες επιφυλάξεις. Έχω επιφυλάξεις σχετικά με την αξία δημιουργίας μιας επιπλέον σήμανσης. Είναι κάτι που είχαμε επισημάνει και στην πρώτη συζήτηση που είχαμε κάνει. Επειδή όμως ο στόχος είναι πάντα η προστασία των καταναλωτών και των πνευματικών δημιουργών, ζητώ τουλάχιστον να μάθουμε από όσα έχουμε πάθει και να αποφύγουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με το σήμα CE. Στο σημείο που η ομάδα μου είχε πρόβλημα να συμφωνήσει είναι το τελευταίο σημείο, το σημείο 8, που έχει να κάνει με την επαναδιάθεση του υλικού που έχει κατασχεθεί ως παραποιημένο παρά τις προϋποθέσεις που προσπάθησε με ειλικρίνεια να θέσει η κυρία Ρόιτοβα και παρά το γεγονός ότι η μέθοδος φαίνεται πως ήδη λειτουργεί σε κάποιες χώρες, ε, φοβόμαστε συγκεκριμένα ότι από τη μια πλευρά μπορεί να ανοίξει ένα παράθυρο να διατίθενται τα προϊόντα αυτά στην αγορά ή να γίνονται ε, αντικείμενα εκμετάλλευσης και από την άλλη πλευρά δεν υπάρχουν εγγυήσεις για την καταλληλότητά του σε σχέση με την ανθρώπινη υγεία. Στο σημείο αυτό επιμένω ιδιαίτερα και καταλαβαίνω ότι και η κυρία Ρόιτοβα ε, είναι γιατρός, έχει ε, θητεύσει υπουργό Υγείας και το καταλαβαίνει και το νιώθει πάρα πολύ καλά, το πιστεύω αυτό. Γι' αυτό τελικά και αν τελικά ε, περάσει η τροπολογία ζητάμε τουλάχιστον ζητώ τουλάχιστον να υπάρχουν εγγυήσει για την ασφάλεια σε σχέση με την υγεία. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ανοχή σας ε, με μία μικρή παρατήρηση. Ότι όταν μιλάμε για επιβολή νομοθεσίας της πνευματικής ιδιοκτησίας μιλάμε για την δικαίωση των δημιουργών. Νομίζω λοιπόν πως είναι πολύ σημαντικό να στηρίξουμε την έρευνα από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης σχετικά με την ίσπραξη και την σωστή διανομή των δικαιωμάτων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ανοχή σας. Δεν ε, είχα σκοπό να ξανανοίξει η συζήτηση. Αυτό θα έπρεπε να είχε γίνει στο παρελθόν ούτως ή άλλως. Ε, τώρα θέλουν και άλλοι το λόγο. Θέλει να απαντήσει και η κυρία Ρόιτοβα. Ε, πρέπει να ψηφίσουμε όμως. Εκτός και αν υπάρχουν λοιπόν θέματα που αφορούν σε ψηφοφορίες ε, και όχι συστάσεις για το πώς να ψηφίσουμε, φαντάζομαι ότι οι πολιτικές ομάδες τα έχουν ήδη κάνει αυτά, να ψηφίσουμε και ε, αργότερα ούτως ή άλλως αυτή η γνωμοδότηση είναι. Θα μπορέσετε να ε, συζητήσετε με την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή και να δείτε πώς μπορείτε να περάσετε τις θέσεις μας. Νομίζω προ τα εκεί θα πρέπει να κατευθύνετε τα πολιτικά σα σχόλια. Νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε τώρα με την ψηφοφορία, εκτό και αν θέλει το λόγο η κυρία Ρόιτοβα. Θέλετε να πείτε κάτι για την ψηφοφορία, λέει ο Πρόεδρο. Ναι. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από την Επιτροπή και την εισηγήτρια. Έκανα λάθος ε, σε αυτά που είπα την προηγούμενη φορά για τις, ε, για τις πιστοποίησεις ήδη υπάρχουν σημάνσεις πιστοποίησης. Ε, τα ε, έμπλεξα αυτά με τις συλλαγικές σημάνσεις και την εθνική νομοθεσία. Συμφωνώ με την κυρία Ρόιτεβα λοιπόν ότι αυτό θα μπορούσε να είναι μια χρήσιμη προσθήκη στην νομοθεσία. Um, Ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Να ψηφίσουμε λοιπόν. Κυρία Ρόιτεβα. Ναι. Έχω μια ερώτηση για την κυρία Ράπτη. Είπατε ότι θα παρουσιάσετε προφορική τροπολογία στην παράγραφο που αφορά στη δυνητική χρήση όταν εκκρεμεί η έγκριση ε, των ε, ε, τσιμάνσεων. Αυτό είπατε στην προφορική σας τροπολογία, διότι ο αρχικός συμβιβασμός ε, ούτως ή άλλως τα ρύθμιζε όλα αυτά, αποσύρθηκε στη συνέχεια ε, κατόπιν δική σα αιτήσεω. Δεν καταλαβαίνω τώρα τι ακριβώ συμβαίνει. Θα συζητήσουμε την προφορική τροπολογία όταν θα φτάσουμε εκεί, λέει ο Πρόεδρο, και έτσι θα είναι πολύ πιο εύκολο να το συζητήσουμε. Δεν... Να διευκολύνω από τώρα, ίσως δεν διατύπωσα σωστά τη σκέψη μου, ε, συμφωνώ με τις, τροπολογι... με, τις ε, με τα κομπρομή, με τους συμβιβασμούς και μόνο αν δεν περάσουν Δηλαδή δεν υπάρχει πρόβλημα. Συμφωνώ με, τις, με τους συμβιβασμούς. Είναι καθαρό τώρα. No, I ε, όχι, αλλά θα το αφήσουμε όταν, για όταν θα φτάσουμε στην ψηφοφορία. Όταν θέλετε να προτείνετε, εάν και εφόσον συγγνώμη, θέλετε να προτείνετε προφορική τροπολογία, θα πρέπει να τη δεχτεί και η Επιτροπή. Θα ήθελα να ζητήσω τώρα από του εισηγητέ και του κοιόδη συζητητέ να προσπαθήσουν να μα οδηγήσουν στην ε, συμβαστική θέση την οποία έχουν συμφωνήσει, εάν την έχουν συμφωνήσει εκ των προτέρων, γιατί αλλιώ ε, δεν θα έπρεπε να επηρεάζουμε την ψηφοφορία. Λοιπόν, τέρμα συζήτηση έχουμε μια νέα ε, παράγραφο μείον 1, τροπολογία 1 της κυρίας του υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται, ε, συντριπτική πλειοψηφία. Συμβιβεστική τροπολογία 1, υπέρ, κατά, δύο κατά, εγκρίνεται και πάλι συντριπτική πλειοψηφία. Να περάσουμε τώρα στην τροπολογία 7, έγκστρομ, υπέρ, να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία μάλλον για την 7. Ε, Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 14 υπέρ 16 κατά. Περνάμε τώρα στη συμβαστική τροπολογία 2. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται και πάλι συντριπτική πλειοψηφία. Να περάσουμε τώρα στην τροπολογία 14 της κυρίας Ρόιτοβα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Παράγραφος 3. Και καταρχήν έχουμε μία τροπολογία του κυρίου Κρόιτσμαν για ε, τη διαγραφή όλης παραγράφου. Υπέρ κατά απορρίπτεται περνάμε τώρα τη συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 3 υπέρ κατά Νομίζω ότι πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικό. Ε, συμβαστική τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε της ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 20 υπέρ 11 κατά. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 20 του κυρίου Μάντερς, υπέρ, κατά, εγκρίνεται, τροπολογία 21 της κυρίας Ρόιτοβα και του κυρίου Έγκστρομ, υπέρ, κατά, εγκρίνεται, συντριπτική και πάλι πλειοψηφία. Συμβιβαστική τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στην τροπολογία 25 του κ. Μάντερς υπέρ. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικώς. Τροπολογία 25. Μάντερς άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 17 υπέρ, 15 κατά. Τροπολογία 26 της κυρίας Τούν υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 27 της κυρίας Ράπτη υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 28 Κρόιτσμαν υπέρ, κατά, Εγκρίνεται συντριπτική και πάλι 29 του κυρίου Μάντερς. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 30. Κρόιτσμαν Άλβαρο. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 31, De Jong, να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ε, τροπολογία 31. Άρχεται η ψηφοφορία. Is... ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 28 υπέρ, 4 κατά. 32 μάντερς υπέρ. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικός. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία του κυρίου σε υπαριθμό 32. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 17 υπέρ 15 κατά. Περνάμε τώρα στη συμβαστική τροπολογία 5 της κυρίας Ρόιτοβα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συντριπτική και πάλι πλειοψηφία. Και τώρα περνάμε στην τροπολογία 37 του κυρίου Μάντερς. Να ε, ψηφίσουμε ηλεκτρονικώς. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 37. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 16 υπέρ, 14 κατά, μία αποχή. Τροπολογία ΣΒΑΜ 38 υπέρ. Α, συγγνώμη, ψηφίζουμε ηλεκτρονικώς. 38 του κυρίου ΣΒΑΜ. Πέραση της ψηφοφορίας εγκρίνεται 17 υπέρ 13 κατά μία αποχή. Τροπολογία 39 Τρασκόφσκι υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 40 του κ. Τρασκόφσκι υπέρ Θα πρέπει να το ελέγξουμε ηλεκτρονικώς. Τροπολογία 40 του κυρίου Τρασκόφσκι. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 16 ψήφοι κατά 14 πέρ. Τροπολογία 41 του κυρίου Τρασκόφσκι. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικώς. Άρχεται η ψηφοφορία. 41 Τρασκόφσκι. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορια ψηφοφορίας. 16-16 απορρίπτεται. Τροπολογία 42 του κ. Τρασκόφσκι. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Να περάσουμε τώρα στη συμβαστική τροπολογία υπερθμών 6. Ρόιτοβα Ντε Υπέρ. Α, συγγνώμη, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικώς. Συμβαστική τροπολογία 6, άρχεται η ψηφοφορία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, πέρες της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 16 ψήφοι υπέρ, 15 κατά, μία αποχή. Και τώρα περνάμε στην επόμενη συμβαστική τροπολογία. Έχουμε, έχει ζητηθεί κατά τμήματα ψηφοφορία για την συμβαστική τροπολογία 7. Επομένως πρέπει απλώς να ελέγξουμε που χωρίζεται. Συμβαστική τροπολογία 7. Uh, Αν κατάλαβα καλά, έχετε ζητήσει κατά τμήματα ε, ψηφοφορία, οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες τη ζήτησαν και ζητούν να χωριστεί ξεχωριστά το τελευταίο τμήμα που λέει emphasize κλπ. κλπ. Ψηφίζουμε ξεχωριστά το κομμάτι αυτό. Προτείνω λοιπόν να ψηφίσουμε πρώτα το πρώτο τμήμα από το encourages μέχρι το counterfeit goods. Ποιοι είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Εγκρίνεται. Και τώρα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικό στο δεύτερο τμήμα Άρχεται η ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα τη συμβαστική τροπολογία 7. Πέρασε ψηφοφορία. Εγκρίνεται 17 ψήφοι υπέρ 14 κατά. Και περνάμε τώρα στην τροπολογία 47. Από μένα. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Δεν υπάρχει καμία ψήφος κατά. Σας ευχαριστώ πολύ. 48. Από τον υποφαινόμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται με συντριπτική πλειοψηφία. Τροπολογία 50 του κυρίου Μάντερ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται και πάλι. 51 της κυρίας Ρόιτοβα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 52 της κυρίας Ρόιτοβα υπέρ, κατά, εγκρίνεται και αυτή. 53 της κυρίας Ρόιτοβα αποσύρεται. The last page. Um, Φτάσαμε στη τελευταία σελίδα. Μπορούμε να ψηφίσουμε όλες αυτές τις ε, ε τροπολογίες σαν blog. Α, όχι, νομίζω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 εγκρίνεται 64 υπέρ. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικώς για την 64. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 19 ψήφι υπέρ 12 κατά. Να περάσουμε τώρα στην τελική ψηφοφορία για το σύνολο της γνωμοδότησης. Ως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 29 ψήφοι υπέρ, 2 κατά και 1 αποχή. Συγχαρητήρια στην κυρία Ρόιτοβα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι τώρα σας περιμένει ενδιαφέρουσα δουλειά με την επί της αρμόδια επιτροπή, την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Να περάσουμε τώρα στην ε, ψηφοφορία για την έκθεση του κυρίου Ρίπο για την ε, πολιτική καινοτομία. Θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Ρέπο. Να ζητήσω από τις κάμερες να απομακρυνθούν λίγο γιατί δεν μπορώ να δω τον κύριο Ρέπο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είχατε δίκιο χθες. Η πρόταση ε, του 3, για το 3% ε, ναι, είναι γεγονός ότι το 3% του ΑΕΠ είναι δημόσια και ιδιωτική ε, επένδυση. Α, ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ γιατί αυτές ήταν και οι στατιστικές που ήξερα εγώ. Άψογα λοιπόν. Ας ε, ξεκινήσουμε λοιπόν την ψηφοφορία για την γνωμοδότηση του κυρίου Ρέπο. Παράγραφος 1, ε, συμβαστική τροπολογία 1, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Επομένως περνάμε στην τροπολογία 3, Κρόιτσμαν, υπέρ, κατά, εγκρίνεται επίσης. Φαίνεται ότι η κυρία Χάιντι Ρούλε θα κάνει μια προφορική τροπολογία. Επομένως ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία της κυρίας Ρούλε ε, σαν ε, προσθήκη υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 3, τροπολογία 5 του εισηγητού, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 5 της κυρίας Ιβάνοβα, υπέρ, κατά 4 ε, συγγνώμη τροπολογία 6 Κρόιτσμαν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 7 τη κυρίας Ιβανόβα υπέρ κατά εγκρίνεται ο τροπολογία 8 Κρόιτσμαν υπέρ κατά εγκρίνεται Τροπολογία 9 Ιβανόβα υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 10 του εισηγητού κυρίου Ρέπο υπέρ κατά εγκρίνεται. Πολύ καλή δουλειά λοιπόν κάνατε κυρία, κύριε Ρέπο και όλοι είναι ευτυχείς με τη δουλειά σας. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά επί του συνόλου. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται λοιπόν μονάχα με μία ψήφο κατά και δύο αποχές. Συγχαρητήρια για την πρώτη σας έκθεση κύριε Σιγητά και είμαι βέβαιος ότι πρόκειται για την πρώτη ε, μιας μακράς σειράς ε, εκθέσεων. Έχουμε τώρα την ε, γνωμοδότηση της κυρίας Μπάστος σχετικά με ψευδεπίγραφα φάρμακα και φαρμακευτικά σκευάσματα. Φαίνεται ότι αγνοείται η τύχη της εισηγητρίας. Έχουμε λοιπόν αγνοούμενο εισηγητή, λέει ο Πρόεδρος. Ε, μπορούμε να μάθουμε αν η κυρία Μπάστος έρχεται, έχει ξεκινήσει.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 Όσο περιμένουμε την κυρία Μπάστος, ας μιλήσει εκ μέρους της ε, Μπάρμπαρα Βάιλερ, σκιώδους εισηγήτριας. Τροπολογίες 23 και 24 αποσύρονται εκ μέρους της ομάδας μου και η κυρία Μπάστος θα παρουσιάσει μια προφορική τροπολογία εν συνεχεία την οποία θα υπερψηφίσουμε. Το λέω αυτό εκ των προτέρων για να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Επίσης, τροπολογίες 18, 37 και 44 της κυρίας Μπάστος τις υποστηρίζουμε. Um, uh, Μήπως κάποιος από τους άλλους σκιώδης ηγητές ε, θέλουν να πάρουν το λόγο πριν ε, έρθει η κυρία Μπάστος για να μην χάσουμε καθόλου χρόνο. Επίσης, ξεκινήσουμε. Έχουμε τη συμβαστική τροπολογία 1 από τους τέσσερις ε, σκιώδεις υπέρ, κατά, εγκρίνονται. Τροπολογία 32 Fox υπέρ. Νομίζω ότι θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 32 Fox άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 23 ψήφοι υπέρ, 10 ψήφοι κατά. 34 και 33 έχουν αποσυρθεί. Τροπολογία 35 Βάιλαρ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία θα κάνουμε. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Κατεψηφίστε 13 ψήφοι υπέρ 19 κατά. Τροπολογία 37 της κυρίας Μπάστος, η οποία βρίσκεται τώρα μεταξύ μας. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η εισηγήτρια είναι εδώ. Ξεκινήσαμε την ψηφοφορία γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Η κυρία Γκέπχαρτ αναφέρθηκε σε κάποια στοιχεία. Μήπως θέλετε εσείς ε, να κάνετε κάποια σχόλια. Σταματάμε λοιπόν την ψηφοφορία για να κάνετε τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ πολύ, ε, Πρόεδρε. Ήμουν ε, σε άλλες ψηφοφορίες στην Επιτροπή Απασχόλησης. Σε πάση περιπτώσει, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις συγητές, καθώς επίσης και όλους τους συναδέλφους που υπέβαλαν τροπολογίες και που μας βοήθησαν μέσω της συνεργασίας τους αυτής να φτάσουμε σε ένα ακόμα πιο θετικό αποτέλεσμα. Ακόμα πιο θετικό λέγω από αυτό που προσδοκούσα μονάχα με την δικιά μου προσπάθεια. Ε, εμπλουτίστηκε λοιπόν η προσπάθειά μου με την συνεργασία όλων και θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους. Βεβαίως το θέμα είναι ε, πολύ ευαίσθητο. Αυτή η πρόταση οδηγίας αφορά ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα και επίσης εδώ αναφέρεται ε, και μία ε, πρωτοβουλία, νομοθετική πρωτοβουλία όσον αφορά τα ψευδεπίγραφα φάρμακα. Γίνεται λόγος για το εμπόριο των ψευδεπίγραφων φαρμάκων και πρέπει να πω ότι η προστασία των χρηστών ε, ασθενών αλλά και η προστασία της βιομηχανίας απέναντι ε, στα ψευδεπίγραφα φάρμακα είναι μέλημα της Επιτροπής μας και την προστασία, τον στόχο αυτό της διτής προστασίας μπορούμε να τον επιτύχουμε ε, με τις προτάσεις μας. Ελπίζω ότι ε, και ε, η, στην τελική ψηφοφορία της Επιτροπής Περιβάλλοντος θα αντικατοπτριστεί η άποψή μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε λέει ο Πρόεδρος. Επομένως, να σας υπενθυμίσω ότι μόλις εγκρίναμε την τροπολογία 37 και επομένως περνάμε στην τροπολογία 36 της κυρίας Βάιλερ. Υπέρ της τροπολογίας 36 Βάιλερ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 39 του κύριου Φόξ έχει αποσυρθεί και επομένως έχουμε τροπολογίες 40 και 41 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 42 της κυρίας Βάιλερ. Νομίζω ότι θα κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία επί της τροπολογίας 42 της κυρίας Βάιλερ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται 17 ψήφι υπέρ 16 κατά μία αποχή. Έχουμε τώρα προφορική τροπολογία της κυρίας Βάστος. Επομένως ψηφίζουμε πρώτα την προφορική τροπολογία της κυρίας Βάστος υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Επομένως η 43 καταπίπτει. Τροπολογία 44 της κυρίας Μπάστος υπέρ κατά εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 6 της κυρίας Μπάστος υπέρ κατά εγκρίνεται. Και επομένως καταπίπτει η 6. Τροπολογία 45 και 46. Α, όχι, όχι, όχι. Δεν χρειάζεται. Επομένως, περνάμε τώρα στην τροπολογία 47. Γιατί η 45 καταπίπτει έτσι κι αλλιώς. Όχι, όχι, πρέπει να ψηφίσουμε επί των 45 και 46. 45 και 46 λοιπόν πρέπει να ψηφίσουμε. Υπέρ, υπέρ των 45 και 46, κατά, νομίζω ότι θα πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Παρακαλώ. Ψηφίζουμε επί των 45 και 46. Ναι, ναι, ε, μπερδεύτηκα λίγο, λέει ο Πρόεδρος. Σύμφωνα με την άποψή μου, δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε για τις 45 και 46, γιατί θα έπρεπε να ψηφίσουμε μονάχα εάν η προφορική τροπολογία της κυρίας Πάστος απερίπτετο. Δεν απερίφθη όμως, πέρασε. Άρα δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Πάστος. Σχετικά με την τροπολογία 47, λέει η κυρία Μπάστο θα ήθελα να καταθέσω προφορική τροπολογία επί του δεύτερου τμήματος. Εκεί δηλαδή που γίνεται λόγος για την εφαρμογή και τα λοιπά, να ληφθεί υπόψη σε ραπρία κονσιντερασιόν. Excuse me. Sorry, I and be linked to the price of the medicinal product concerned passa a ser should μετά το concern δηλαδή να πούμε medicinal products will be κτλ. Α, αναφέρεσαι στην τιμή λέει ο πρόεδρος. Ναι. Ναι, should take into consideration the price of the medicine. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η τιμή του φαρμάκου. Okay. Okay. Uh, right. Thank you. Okay. Can I just clarify? Because I was asked... Λοιπόν, η, η ουσία είναι ότι εγώ μιλούσα εκείνη την ώρα για τις τροπολογίες 45 και 46 ε, και αποφασίσαμε ότι τελικά δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε από τον 45 και 46. Επομένως τώρα φτάνουμε ε, στην τροπολογία 47. Προτρέξατε λίγο, δεν πειράζει. Εδώ έχουμε χωριστή ψηφοφορία επί της ε, τροπολογίας 47 της κυρίας Παρβάνοβα να ξεκινήσουμε με ψηφοφορία επί του πρώτου τμήματος και μετά να συνεχίσουμε. Υπέρ του πρώτου τμήματος της 47, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Έχουμε τώρα το δεύτερο τμήμα και η κυρία Μπάστος προτείνει προφορική τροπολογία που να λέει λοιπόν ότι θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την τιμή της, ε, του, του ε, φαρμάκου. Και η κυρία Παρβανόβα συμφωνεί, επομένως υπέρ, κατά, η προφορική τροπολογία γίνεται δεκτή. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 7. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 49 48 του κυρίου Φόξ υπέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία 49 Βάιλερ υπέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία 50 Βάιλερ υπέρ κατά εγκρίνεται Τροπολογία 8 μπάστος υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 9 μπάστος υπέρ κατά απο, εγκρίνεται. Τροπολογία 51 παρβάνοβα υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 52 Βάιλερ υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 10 Μπάστος υπέρ κατά εγκρίνεται επίσης. Άρθρο 2, τροπολογία 53, Fox. Άρχεται η ψηφοφορία, θα κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 53 του κυρίου Fox. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται λοιπόν 23 ψήφοι πέρα 11 κατά. Τροπολογία 54 του κυρίου Φόξ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 54 πέρας της ψηφοφορίας ε, δεκτή 25 προς 9 55 του κυρίου Φόξ άρχεται ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας δεκτή 22 προς 11 τροπολογία 56 την ψηφίζουμε ρωτάει ο πρόεδρος 56 καταπίπτει, διότι διεχτήκαμε την 32. Τώρα προχωρούμε στα εκτιμώντα. Τροπολογία 11, Μάντερς. Άρχεται η ψηφοφορία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ε, τροπολογία 1 έχει αποσυρθεί. 13, κυρίες Μπάστος. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται. Άρχεται. Τροπολογία 13 είμαστε. πέρα τη ψηφοφορία. Δεκτή. 22 προς 11. Οπότε καταπίπτει τροπολογία 12. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Α, αποχές δεκτή. 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 17. Υπέρ κατά, αποχές δεκτή, 19 έχει αποσυρθεί, 18 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, 3, τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, 20 και 21 υπέρ, κατά, απορρίπτεται, απορρίπτονται, Ψηφίζουμε την 22. Ψηφίζουμε την 22 υπέρ, κατά, άποχες, ε, απορρίπτεται. 20-24 απεσύρθησαν μαζί με την 25, προχωρούμε στην 26 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή και τέλος Τροπολογία 27, Παρβάνοβα, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τώρα ψηφίζουμε την, ε, το σχέδιο γνωμοδότησης. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 32 υπέρ με δύο εποχές. Συγχαρητήρια κυρία Μπάστος. Σας ευχαριστούμε. Ευχόμαστε σε εσά και, στην, και στους χειώδεις εισηγητές κάθε επιτυχία. σύντομο διάλειμμα μέχρι τις 11 και θα συνεχίσουμε με την έκθεση της κυρίας Σουρίντο. Κοιτούσα uh, απλώ να δω αν είναι ο εκπρόσωπο τη Επιτροπή εδώ. Θα έρθει. Είναι καθοδόν. Θέλετε να τον περιμένουμε. Uh, Νομίζω λοιπόν Μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, διότι έχουμε μία ε, πάρα πολύ μεγάλη έκθεση από την κυρία Ρούλε. Δεν ξέρω αν είναι εδώ όλοι οι σκιώδεις συγητές. Έχουμε κάτι λήψη σε σκιώδεις. Ο κύριος Έγγελ είναι εδώ. Μπορεί να χρειαστεί ίσως να περιμένουμε να έρθουν όλοι οι σκιώδεις συγητές. Ο κύριος Κρότσμεν είναι εδώ, εγώ είμαι εδώ. Ο κύριος τρενταφυλλιδης είναι εδώ. Ε, λείπουν όμως ένα-δυο συνάδελφοι. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο, αν δεν σας πειράζει. Ο κύριος Έγγελ θα έρθει. Ο κύριος Έγγελ και η κυρία Βένιου πρέπει να έρθουν γιατί χρειάζεστε και τους κοιόδης συζητητές για αυτή τη συζήτηση. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ομάδα των σκιο... σκιωδών εισηγητών είναι εδώ εν απαρτία. ο κύριος Βίνο έρχεται επίση. Και επίση έχουμε εδώ τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, τη Γενική Διεύθυνση και έτσι μπορούμε να αρχίσουμε και δίνω το λόγο στην κυρία Ρούλε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ήδη έχω συζητήσει με την Κομισιόν το θέμα αυτό, οπότε μια μικρή καθυστέρηση δεν δημιουργεί πρόβλημα. Ευχαριστώ τους και τους για την εμπιστοσύνη τους και την καλή συνεργασία. Και ελπίζω να μην τους απογοήτευσα και ειδικά ευχαριστώ τη Γραμματεία για το περιθώριο ελιγμού το οποίο μου έδωσαν. Συνήθως ε, θα μου δίναν τέσσερις σελίδες, αλλά φρόντισα να πάρω λίγο περισσότερο χώρο και ευχαριστώ ιδιαίτερα. Είναι ένα πολύ πυκνό και συμπιεσμένο κείμενο. Έχω η ίδια υποβάλει τροπολογίες. Έχω στείλει τα στοιχεία σε όλους όσους θέλουν να υποβάλουν. Έχω αλλάξει τη δομή της ε, έκθεσης διότι έχω τώρα περισσότερο χώρο με τις τροπολογίες και έτσι μπορεί το κείμενο να γίνει πιο κατανοητό και να έχει περισσότερη πολιτική ισχύ. Θα στείλω λοιπόν τη νέα δομή του κειμένου πάρα πολύ σύντομα, όσο πιο σύντομα μπορώ, ήθελα απλώς να σας ε, το διευκρινίσω. Βεβαίως ε, είναι ένα συμβιβαστικό κείμενο, συμπιεσμένο, δεν είχαμε πάρα πολύ καιρό αλλά συζήτησα με την πρακτική πλευρά, με τους πρακτικά ενδιαφερόμενους από, τον, από την οικονομική πλευρά, από τη βιομηχανική πλευρά, από την πλευρά του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ρώτησα ποια είναι τα προβλήματα. Δεν μπόρεσα να καταγράψω και να καλύψω όλα τα προβλήματα, παραδείγματο χάρη κοινωνικέ κατοικίε. το θέμα των εργατικών όπω λέμε εμεί, κατοικιών, δηλαδή κατοικιών που χτίζονται από το δημόσιο. Ε, αυτά όλα είναι θέματα της πολεοδομία και της χωροταξίας και βλέπουμε ότι στι δημόσιε συμβάσει υπάρχει πάρα πολύ πυκνή νομοθεσία. Κανόνες επί κανόνων και νόμοι επί νόμων κανονισμούς και τα λοιπά και τελικά οι τοπικές αρχές, η τοπική αυτοδιοίκηση περιορίζεται εξαιρετικά από αυτή την κεντρική νομοθεσία. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και διαφορετικές ερμηνείες από τα εθνικά δικαστήρια έναντι του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Υπάρχουν τώρα καταστάσεις που έχουν προκύψει που από τον νομοθέτη δεν το σκέφτηκε ποτέ. Παραδείγματος χάρη η πώληση οικοπαίδων ε, ανήκει στο δημόσιο τομέα. Σήμερα όμως όταν η κοινότητα πουλάει κόπεδα, τα πουλάει επειδή θέλει να εφαρμόσει μία στεγαστική πολιτική Παραδείγματο χάρη, αν θέλει να προσελκύσει επιχειρήσεις, πουλάει ένα οικόπεδο σε μια εταιρεία πληροφορικής, οπότε θεωρείται αυτή η πώληση, ε, πώληση προστιθέμενης αξίας. Άρα εμπίπτει στις διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων κατά τη γερμανική νομοθεσία. Άρα λοιπόν οι δημόσιες συμβάσεις δεν περιορίζονται μόνο σε τομείς τους οποίους καλύπτει η νομοθεσία. Έχουν προκύψει άλλες δυνατότητες και άλλες ερμηνείες τις οποίες τώρα πρέπει να καλύψουμε που δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Αλλά βεβαίως λόγω του πολύ πυκνού νομοθετικού πλαισίου η ευελιξία είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Θέλω να παρακαλέσω την Κομισιό να εξετάσει ε, εις βάθος αυτή την πρόταση, να εξετάσει όλες τις πτυχές αυτού του ευρύτατου τομέα. Ιδίως οι πτυχές που αναφέρονται σύντομα στην έκθεσή μας. Όταν στην, στον κατασκευαστικό τομέα υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ Ευρωπαϊκών ευρωπαϊκών εταιριών και μη ευρωπαϊκών εταιριών οι οποίες επιδοτούνται από τις κυβερνήσεις τους. Αυτοί είναι τομείς που δεν εμπίπτουν στο δικό μου θέμα, δηλαδή ανταγωνισμός μεταξύ κοινότητα Ευρωπαϊκής Ένωσης και εταιριών που επιδοτούνται από τρίτες χώρες. Αυτό δεν μπορούσα να το καλύψω, αλλά η Κομισιόν θα ήθελα να τα εξετάσει όλα. Αυτό που εγώ επιδιώκω είναι δημιουργία νομικής ασφάλειας και η ενθάρρυνση του δημόσιου τομέα να μην ε, δέχεται πάντοτε τη φτηνότερη σύμβαση σε έναν μειοδοτικό διαγωνισμό, αλλά να, έχει τη δυνατότητα να δέχεται την καλύτερη πρόταση, την καλύτερη σύμβαση. Ε, επειδή υπάρχει στενότητα οικονομική αλλά και νομική ανασφάλεια, συνήθως γίνονται δεκτές οι φθηνότερες προσφορές που δεν είναι πάντα οι καλύτερες. Γι' αυτό παρακαλώ την Κομισιόν να παράσχει περισσότερη βοήθεια, περισσότερη ενίσχυση, καλύτερο συντονισμό και καλύτερη διεύθυνση, καλύτερη ηγεσία, έτσι ώστε η Γενική Διεύθυνση που είναι η επί της ουσίας ε, αρμόδια να αναλάβει τις ευθύνες της για έναν θεμητό ανταγωνισμό. έτσι ώστε και οι ανασέτοντες αλλά και οι συμβασιούχοι να μπορούν να αναγνωρίσουν, αυτοί που παίρνουν δηλαδή τα συμβάσεις, ε, οι δικαιούχοι να μπορούν να αναγνωρίσουν ακριβώς τους κανόνες του παιχνιδιού. Οι κανόνες του παιχνιδιού σε, πολλές, ε, σε πολλούς τομείς είναι ασαφείς, είναι μπερδεμένοι ε, και η πρόταση αυτή έχει δημιουργήσει πολλά επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα δεν είναι σωστό να δεχόμαστε πάντοτε την φτηνότερη προσφορά. Ε, φτύνια ή ποιότητα. Πρέπει να έχουμε μία ευελιξία. Να μην στριμωχνόμαστε και να μας οδηγεί πάντοτε η επιλογή μας προς το χαμηλότερο κόστος, το φτηνότερο. Να έχουμε την ευελιξία επιλογής ποιότητος. τη Γερμανία, παραδείγματος χάρη, Ε, ακούγονται πολλές επικρίσεις για το πώς ρυθμίζεται στη Γερμανία η ανάθεση συμβάσεων. Για την ανάθεση, την πλευρά της ανάθεσης υπάρχουν πολλές επικρίσεις, υπάρχει ασάφεια, δεν υπάρχει νομική ασφάλεια και αυτά θέλω να διορθωθούν. Και τέλος υπήρχε και ασάφεια ε, ε, από πλευράς μεταφράσεων. Η γαλλική μετάφραση ε, έχει μεταφράσει το δημόσιο ως δημόσιο ιδιωτικό. Ε, επίσης υπάρχει ασάφεια ε, στις, στους ορισμούς και στις μεταφράσεις τους. Παρακαλώ λοιπόν να λυθούν τα μεταφραστικά προβλήματα. Έχω ήδη διορθώσει την αγγλική έκδοση και έχω αποφασίσει να εργαστώ επί της αγγλικής μετάφρασης, όχι της γερμανικής, διότι περιέχει πολλά λάθη. Αυτά είχα να πω ε, αρχικά. Ελπίζω να καταλήξουμε σε μια ισχυρή υπερψηφία. Α, και κάτι άλλο, να μην ξεχάσω. Νέα νομοθεσία, καινούργια νομοθεσία. Όλοι ξέρετε ότι η Κομισιόν έχει αναθέσει ε, μελέτη στο θέμα της παροχής υπηρεσιών, σε αυτό τον τομέα. Προσωπικά έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είναι λάθος σήμερα να υιοθετήσουμε νέες νομοθετικές ρυθμίσεις πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να περιμένουμε την αξιολόγηση της Κομισιόν η οποία θα πρέπει να εξετάσει εις βάθος την ε, οδηγία του νομικού πλαισίου παροχής υπηρεσιών και να μην προτείνει η Κομισιόν νέα νομοθεσία πριν περάσουν δύο-τρία χρόνια και παγιωθεί η υπάρχουσα νομοθεσία και αξιολογηθεί. Συζήτησα με εκπροσώπους από όλα τα κράτη-μέλη, συζήτησα με τοπικές αυτοδιοικήσεις και με επιχειρήσεις και με παρακάλεσαν όλοι οι φορείς να μην τους ε, επιβαρύνουμε με περισσότερη νομοθεσία διότι θα στριμωχτούν ακόμα περισσότερο, θα δεσμευτούν και δεν θα έχουν πια καθόλου ευελιξία οι αναθέσεις στον τομέα των υπηρεσιών, οι, οι και οι όλες οι ρυθμίσεις του τομέα των υπηρεσιών στα κράτη-μέλη είναι διαφορετικές. Δεν το αμφισβητώ, όμως δεν πιστεύω ότι δημιουργούν σοβαρές τρευλώσεις της αγοράς. Δεν έχουμε τέτοιες αποδείξεις τουλάχιστον. Γι' αυτό προ όφελο των δημοσίων αναθέσεων δεν θα ήθελα να προβάλλει η Κομισιόν περαιτέρω νομοθετικές προτάσεις πριν περάσουν αυτά τα δύο-τρία χρόνια της παγίωσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Ρίλε για την ε, πολύ εμπεριστατωμένη έκθεση την οποία θα εξετάσω λεπτομερώς ο, ο πρόεδρος ε, δίνει την άδεια των ε, περισσότερων σελίδων. Ε, η γραμματεία απλώς εγκρίνει την πρόταση του πρόεδρου. Δεν δίνω αυτό το δικαίωμα σε όλους, αλλά σε εσά το έδωσα να έχετε λίγο περισσότερο χώρο στο κείμενο. Έχουμε ε, ένα ισχυρό, μια ισχυρή ομάδα εκπροσώπων της Κομισιόν από τη Γενική Διεύθυνση ε, Εσωτερικής Αγοράς και επίσης έχουμε και τη συνάδελφό μας από την ε, Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων και, και την κυρία Ντεγκρού η οποία έχει αναλάβει την πράσινη κάρτα την οποία προηγουμένως στο παρελθόν είχε ο κύριος Μπαλνιέ. Καταρχάς δίνω το λόγο στους κοιόδης εισηγητές. Α, κύριε Χάνσλερ, κύριε Γκέπαρτ. Και εγώ είμαι σκιώδης. Ο κύριος Τοιανταφυλλίδης, η κυρία Γκέπαρτ. Ο κύριος Σβάμπ καταρχάς. Ε, Άλλο ομιλητής, ομιλήτρια, κύριε Σφαμπ. Ναι, Ωραία. Έχουμε λοιπόν άνεση χρόνου, αλλά θα να δώσω και το λόγο στην Κομισιόν. Ε, ο κύριος Έγκελ έχει το λόγο καταρχάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω υπογραμμίζοντας όπως και εσείς άλλωστε την ε, εξαιρετική ποιότητα της ε, έκθεσης κυρίας Ρούλε και να την ευχαριστήσω επίσης για την πάντα διαθέσιμη για οποιαδήποτε συνεργασία ή αποτελεσματική ανταλλαγή απόψεων. Χαιρετίζω σε αυτό το δύσκολο τομέα την επιλογή της εισηγήτριας να υπογραμμίσει κυρίως την ανάγκη αύξησης της ασφαλείας δικαίου σε ένα τομέα ο οποίος δεν μπορεί να θεσμοθετηθεί ε, πλήρως γιατί θα, αυτό θα οδηγούσε σε στρεβλώσεις. Είναι ένας κλάδος βεβαίως ε, στον οποίο πάντα θα βρεθεί αυτός ο οποίος θα πει ότι ζημιώνεται με τις νέες ε, διατάξεις. Όμως αυτό δεν μας εμποδίζει από το να πούμε σαφώς ότι θα πρέπει να αυξήσουμε την ασφάλεια η οποία πρέπει και μπορεί να υπάρχει και επομένως να διευκολύνουμε ε, αυτό, ε, το έργο αυτών των ανδρών και γυναικών που καλούνται να πάρουν τις τελικές αποφάσεις όσον αφορά την, ε, την τελική επιλογή για τις δημόσιες συμβάσεις. Στον τομέα αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα δικαιώματα και αυτών που ε, προτίθενται να υπογράψουν συμβάσεις ε, και αυτών που προτείνουν τις συμβάσεις. Ε, βεβαίως, το καλύτερο κριτήριο, κυρίως σε σχέση και με το νέο, ας το πούμε, εντό αγωγικών κριτήριο, το, το, των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι η καλύτερη προσφορά, η μικρότερη δηλαδή οικονομική ε, προσφορά. Αυτό είναι ε, ο κανόνας όσον αφορά τις ε, δημόσιες συμβάσεις. και επομένως ε, θα πρέπει να δημιουργηθούν ε, οι προϋποθέσεις αυτές ε, οι οποίες θα επιτρέπουν να είναι τελικά και η πιο σωστή επιλογή αυτή της προσφοράς που είναι πιο συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως. συνδυασμού πάντα με τα καινούργια αυτά κριτήρια. Βεβαίως είναι γεγονός ότι οι δημόσιες ε, συμβάσεις είναι κάτι που απασχολεί όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου. Ε, πρέπει όμως ε, να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας. Επίσης, όσον αφορά την παροχή... Όσον αφορά τις εκχωρήσεις υπηρεσιών, θα συμφωνήσω και εδώ με την κυρία Ρούλε, δηλαδή ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ε, δηλαδή να μην προσπαθήσουμε οπωσδήποτε να επιβάλλουμε ε, διατάξεις ε, παραμονάχα εάν πραγματικά βλέπουμε στρέβλωση του ανταγωνισμού ή της αγοράς. Εάν η Κομισιόν θέλει να προχωρήσει νομικές διατάξεις όσον αφορά τις παραχωρήσεις δικαιωμάτων παροχής υπηρεσιών, τότε θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει αποσαφήνιση ε, για το πεδίο εφαρμογής, ε, δηλαδή τι θα πρέπει ε, να διευκρινιστεί, τι θα πρέπει να διευθετηθεί γιατί εμείς είχαμε υποβάλει και επί του προκειμένου διάφορα ερωτήματα τα οποία ποτέ δεν απαντήθηκαν. εμείς αυτό που θέλουμε να ξέρουμε είναι εάν θα νομοθετήσουμε όσον αφορά το θέμα αυτό και αν ναι μέχρι ποιο βαθμό. Ποτέ δεν είχαμε σαφή απάντηση. Ολοκληρώνοντας κύριε Πρόεδρε, και αυτή είναι και μία από τις προτάσεις ε, που έχω συγκρατήσει και από το δικό μου κράτος, ε, που είναι και μάλιστα πολύ μικρό κράτος. Φαίνεται ότι δεν θέλουν ούτε περισσότερη ούτε νέα νομοθεσία οι εμπλεκόμενοι φορείς. και νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο η κυρία Ρούλε απαντάει ε, στο αίτημα, πούμε, στην επιθυμία αυτή. Ε, δηλαδή να μην κάνουμε υπερβολική νομοθεσία, να νομοθετήσουμε εκεί που είναι απαραίτητο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Χάιντε Ρούλε για την εξαίρετη ε, εργασία της αλλά και για το ευρύ πνεύμα συνεργασίας το οποίο έχει επιδείξει γιατί πραγματικά έλαβε υπόψη της ε, όλες τις επιθυμίες ε, και τα σχόλια των σκιωδών εισηγητών στις συναντήσεις που έκανε μαζί μας. Σημερίζομαι την άποψή της ε, δηλαδή ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να αρθεί η νομική αβεβαιότητα όσον αφορά τα θέματα αυτά. Ε, αβεβαιότητα η οποία είναι ζημιογόνα και όσον αφορά τους υπεύθυνους των δημοσίων συμβάσεων και όσον αφορά τις επιχειρήσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εδώ έχουμε ε, μία σειρά πρωτοβουλειών που μερικές φορές αντιτίθενται η μία στην άλλη και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν ήδη αποδοκιμαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Έχουμε ήδη αρνητικές ε, ετοιμιγορίες όσον αφορά τις συμπράξεις ε, δημοσίου και ιδιωτικού. Εν πάση περιπτώσει ελπίζω ότι οι υπεύθυνοι της Επιτροπής ε, θα λάβουν υπόψη όλα τα στοιχεία αυτά έτσι ώστε ε, χωρίς να κάνουμε επιπλέον νομοθέτηση να ε, υπάρξει περαιτέρω αποσαφήνιση ε, των ελληπών διατάξεων. Χρειαζόμαστε νομική διασαφήνιση για όλα αυτά τα θέματα. Υπάρχουν ακόμα και κάποια θέματα, κάποια σημεία τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να ξανασυζητηθούν όσον αφορά ε, την πολεοδομία και όσον αφορά τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Πιστεύω ότι εδώ θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε τα σημεία αυτά. Θα πρέπει να επιφέρουμε διευκρινήσεις, κυρίως όσον αφορά τις κοινωνικές ρήτρες. Ε, αναφέρομαι ας πούμε σε χώρες όπου ε, αναφερόμαστε κυρίως σε νέους έφηβους καμιά φορά εργαζόμενους, ε, εργαζόμενους με προβλήματα αναπηρίας κτλ. Εδώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα εισαγωγής τέτοιου είδους κριτηρίων τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το κοινωνικό και περιβαλλοντικό μοντέλο το οποίο όλοι μας αναφέραμε και του οποίου όλοι μας υπεραμεινθήκαμε στην τελευταία προεκλογική εκστρατεία. Πιστεύω ότι θα πρέπει και μέσω αυτών των στοιχείων να δώσουμε περισσότερη εμπιστοσύνη ε, στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα και βεβαίω δεν είναι δυνατόν το μόνο κριτήριο να είναι η, η χαμηλότερη τιμή, αλλά η καλύτερη τιμή. Η καλύτερη τιμή δηλαδή μια τιμή λογική, η οποία όμως θα ε, αναφέρεται και σε όλα αυτά τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά στοιχεία τα οποία αναφέραμε προηγουμένως. Τελευταία σύντομη παρατήρηση. Συμφωνώ απολύτως ε, με την εισηγήτρια όσον αφορά τα προβλήματα μετάφρασης των τροπολογιών. Μερικές φορές είναι εξαιρετικά ενοχλητική η κατάσταση. Θα ζητήσω από τη Γραμματεία να επιληφθεί του θέματος. Να δώσουμε και κάποια παραδείγματα, ίσως θα βοηθήσουμε έτσι. Ο κύριος Κρόιτσμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ με τη σειρά μου θα πρέπει να ευχαριστήσω την κυρία Ρούλε, η οποία έκανε εξαιρετική δουλειά και η οποία αναφέρθηκε κυρίως ε, στη συνεργασία ε, για το θέμα το οποίο συζητούμε. Σήμερα το πρωί μιλήσαμε για την πιο ευνοϊκή ε, προσφορά από οικονομικής πλευράς ή την πιο φθηνή προσφορά. Προσέξτε, δεν είναι πάντα το ίδιο πράγμα αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχουν ανταγωνιστές ε, στις δημόσιες συμβάσεις, να δίνονται ίσες ευκαιρίες στις ιδιωτικές επιχειρήσεις για να μπορούν να συμμετάσχουν. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην ε, ε κίνηση γειτονίες ε, ανοίξαμε τις δημόσιες συμβάσεις ε, και στις τοπικές αρχές. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα πρέπει να είναι οι ομοσπονδιακοί σιδηράδρομοι αυτοί οι οποίοι θα κερδίζουν τους δημόσιους ε, διαγωνισμούς και θα λαμβάνουν την εντολή να εκπονήσουν το έργο. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιος ανταγωνισμός. Και πρέπει να πω ότι τα ομόσπονδα κρατήδια τελικά εκχώρησαν δημόσιες συμβάσεις Τελικά ε, ο διαγωνισμός ε, ε, δόθηκε στην Bundesbank αλλά όχι γιατί ήταν η μόνη η οποία έκανε την προσφορά αλλά γιατί έκανε την πιο οικονομική προσφορά. Επιτρέψτε μου λοιπόν να παρουσιάσω μια τροπολογία η οποία λέει ότι οι δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να είναι και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για να υπάρχει και ανταγωνισμός επί ίσης όρης. Θα ήθελα επίσης να σταθώ και στα οικολογικά και κοινωνικά κριτήρια. Σαφώς θα πρέπει και αυτά τα στοιχεία να λαμβάνονται υπόψη σε ένα μειοδοτικό διαγωνισμό για να μην οδηγηθούμε και σε καταστάσεις ε, οι οποίες δεν θα λαμβάνουν υπόψη, ε, για παράδειγμα, ε, μια επιχείρηση ε, στην οποία εργάζονται άτομα με αναπηρία. Αυτό ε, γίνεται στη Γερμανία για να λάβουμε υπόψη και θέματα κοινωνική ευθύνη. Αλλιώ δεν του δίνονται ίσες ευκαιρίε ανταγωνισμού στην αγορά. Ε, αυτά τα κριτήρια θα πρέπει να λαμβάνονται κατά κάποιο τρόπο υπόψη από πλευρά όσων εξετάζουν φακέλου συμμετοχή σε μειοδοτικού διαγωνισμού. Επίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ετοιμάσουν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, κάποιους προσανατολισμούς ώστε η νομοθεσία να ε, μπορεί να οδηγήσει και σε κάποια πράγματα σε τοπικό, σε περιφερειακό επίπεδο. Δεδομένου ότι οι τοπικές αρχές πολλές φορές ε, είναι υπερβολικά φορτωμένες και για να μπορούν να έχουν και οι τοπικοί φορείς τη δυνατότητα να αντιδράσουν, να κρίνουν. Ευχαριστούμε λοιπόν την εισηγήτρια και πιστεύω ότι θα τύχουμε της πλειοψηφίας εδώ. Θα υπάρχει πλειοψηφία. Ο Πρόεδρος. Επιτρέψτε μου να ε, μιλήσω κι εγώ λίγο, να κλέψω λίγο από τη λάμψη σα, διότι κι εγώ είμαι σκιώδη εισηγητή στο θέμα αυτό. Ήδη στην την κυρία Ρούλα για την προσέγγιση που ακολούθησε σε αυτή την έκθεση. Θα ήθελα να κάνω και κάποια γενικά σχόλια, γενικώ για τι δημόσιε συμβάσει τα οποία ίσως αντικατοπτρίζουν και την στάση μου για την έκθεση αυτή. Όταν επισκέπτομαι δημόσιες αρχές διαπιστώνω ότι σε πολλές περιπτώσεις το σύνολο του καθεστώτος δημοσίων συμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρείται ως κάτι ε, γραφειοκρατικό, μία όχληση που δεν ε, ευνοεί απαραίτητα τις συνθήκες εργασίας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, πρόβλημα αντίληψης. Θα πρέπει να πούμε λοιπόν και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει ίσως να διορθώσουμε. Θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε και με την κυρία Ρέντινγκ που ήταν εδώ εχθές, ε, η οποία είναι υπεύθυνη για τα θέματα επικοινωνίας ε, σε αυτή την περίπτωση. Όπως βλέπουμε και στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020, είναι πάρα πολύ σημαντική η στρατηγική χρήση των δημόσιων συμβάσεων. Αυτό θα αποτελέσει ένα βασικό μέσο για να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε ε, κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική μεταρρύθμιση. Θα βοηθήσουμε τον ανταγωνισμό και θα συνδράμουμε και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ε, δεν συζητούμε όμως με τις τοπικές αρχές για το πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτό το μέσο με ρεαλιστικό και λογικό τρόπο. Και επίσης φρονώ ότι πολλά από τα γραφειοκρατικά θέματα ίσως ε, υπερβάλλουμε όταν τα αναφέρουμε γιατί τίνουμε να κάνουμε τη ζωή μας πολύ πιο περίπλοκη. Οι δημόσιες αρχές θεωρούν ότι θα πρέπει πάντα να μιλήσουμε νομικούς συμβούλους ε, διότι ε, θεωρούν ότι έτσι λειτουργούν τα πράγματα και αυτό αναφέρεται με πολύ περιγραφικό τρόπο στην έκθεση της κυρίας Ρούλε και πολλά πράγματα γίνονται και πολύ πιο περίπλοκα. Πολλές συμβάσεις είναι πιο περίπλοκες. Κάποιες από τις διαδικασίες που ζητούνται να ακολουθηθούν θα πρέπει ε, να εξετάζονται και υπό το πρίσμα του καλύτερου αποτελέσματος. Να μην θεωρούμε ότι είναι απλώς μία ε, επαχθής διαδικασία θα πρέπει να υπάρχει μια ε, διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου που είναι υπέρ και του πελάτη και του ε, δυνητικού προμηθευτή να δώσει κάτι το οποίο ε, θα τηρεί τις βασικές απαιτήσει που θέλει να επιτύχει μια σύμβεση. Έτσι θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και καλύτερη σχέση κόστους-οφελίας. Κάπου όλα αυτά φαίνεται να τα χάνουμε γιατί ε, ασχολούμαστε πιο πολύ με τα νομικά θέματα. Και νομίζω ότι εμείς ως Επιτροπή θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό το θέμα διότι είμαστε υπέρμαχοι των καλύτερων δημοσίων συμβάσεων αλλά καταλαβαίνουμε και τη σημασία των δημοσίων συμβάσεων ως ένα εργαλείο για τη δημόσια πολιτική μας. Υπάρχουν λοιπόν πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και που θα μπορούσαν να είναι πιο αποτελεσματικά και ε, νομίζω ότι θα πρέπει να το λάβουν υπόψη και οι κρατικές αρχές αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τις συμβάσεις αυτή τη στιγμή δεν είναι κατά ανάγκη ο βέλτιστο δυνατός. Ε, αυτά ω προκαταρκτικά σχόλια. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία ανέφεραν και οι συνάδελφοι, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να επισημάνουμε. Είναι το δυνατότητα συμμετοχή σε δημόσιε συμβάσει μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στην πράξη, μια μικρομεσαία επιχείρηση θα πρέπει να θεωρεί τη δημόσια σύμβαση ως μια εξαιρετική ευκαιρία, διότι τους παρέχει πρόσβαση μέσω διαδικτύου σε μια τεράστια βάση δεδομένων ε, συμβάσεων που έχουν ήδη λάβει μια πρώτερη έγκριση, να δουν τι ακριβώς θέλουν, τι ακριβώς θέλουν να ακολουθήσουν και πού μπορούν να αναζητήσουν και αυτοί περαιτέρω εργασία για την επιχείρησή τους. Και για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έπρεπε αυτό να είναι μια εξαιρετική ευκαιρία. Ε, φοβάμαι όμως ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν το βλέπουν έτσι, γιατί ακόμα και για την προκαταρκτική έγκριση ε, θα πρέπει να περάσουν από μια πολύ ε, επώδυνη γραφειοκρατική διαδικασία και σε πολλές περιπτώσεις είναι τόσο περίπλοκες οι διαδικασίες και δεν γίνεται κάποιος κατακαιρματισμός ε, ή δεν υπάρχει κάποια δυνατότητα υπεργολαβίας ε, για να μπορέσουν να συμμετάσχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος είναι μάλλον αυτό στο οποίο θα έπρεπε να εστιάσουμε κάποιοι συνάδελφοι είναι υπέρ κάποιου κατοχλίου, να υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο το οποίο θα δίνεται στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Νομίζω ότι έτσι όμω παρακάμπτουμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι γιατί δεν συμμετέχουν οι μικρομεσαίε επιχειρήσει και ποια είναι τα προσκόμματα που δεν του επιτρέπουν να μπορέσουν να συμμετέχουν σε μια διαδικασία που κανονικά θα έπρεπε να είναι μια ε, μεγάλη πηγή δυνητικής εργασίας για αυτούς ε, έργου. Ε, πολλές ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, τα αποφεύγουν ακριβώς λόγω μεγάλου άχθους. Τέλος να πω κάποια πράγματα για τον ενθουσιασμό μου για τις καινοτόμες συμβάσεις. Αναφέρθηκε και λίγο πριν. Η κυρία Ρούλε είπε στην αρχή ότι θεώρησε ότι το καλύπταμε καταλήλω στην έκθεσή μου του 2008 και με κολακεύει το γεγονός ότι θεωρεί ότι το καλύπτουμε. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή θα μπορούσε να υποφοληθεί αν είχαμε μία σύνοψη των συστάσεων της προηγούμενης έκθεσης. Θα ήταν μια ενίσχυση της εκθέσεως και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά κάποιες από αυτές τις συστάσεις. Ε, στέκομαι κυρίως στο γεγονός ότι οι δομές που απαιτούνται προκειμένου να ενθαρρύνουμε όσους συμμετέχουν σε δημόσιες συμβάσεις να ε, συμπεριφέρονται με πιο καινοτόμο τρόπο ε, αναπτύχθηκαν στην ε, Γενική Διεύθυνση ε, της Κοινωνίας της Πληροφορίας και όχι στη Γενική Διεύθυνση Μάρκτ το θέμα αυτό θα συζητηθεί και πολύ εδώ στις Βρυξέλλες και να σας πω ότι έχω προσκληθεί και σε κάποια διάσκεψη για να μιλήσω γι' αυτό. Θα έχετε λάβει και τα στοιχεία. Αλλά ε, νομίζω ότι πλέον συμμετέχει και η Γενική Διεύθυνση Enterprise. Επομένως έχουμε τρία τμήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασχολούνται με το θέμα. Ε, νομίζω όμως ότι θα πρέπει να το προωθήσουμε ακόμα πιο ενεργά και νομίζω ότι όλα αυτά ενθαρρύνουν όλους όσους ασχολούνται με τις δημόσιες συμβάσεις να τα προσέξουν πολύ περισσότερο, διότι θα υποφοληθούν και οι δύο πλευρές. Θα έχουν καλύτερες και πιο καινοτόμες λύσεις και ταυτόχρονα θα δοθεί μια έθωση στην οικονομία και στις καινοτόμες επιχειρήσεις που θέλουμε να έχουμε αν ε, μου επιτρέψετε λοιπόν να προτείνω κάποια πράγματα εδώ, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να είναι το επίκεντρο της έκθεσης, αλλά καλό θα ήταν να ενισχύσουμε τη δέσμευσή μας επί του θέματος αυτού, κυρίως γιατί αυτή τη στιγμή αναφέρεται ρητός ε, στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020 ως ε, στοιχείο καινοτομία, κάτι που με χαροποιεί ιδιαίτερα και νομίζω ότι θα πρέπει και εμείς να το ενδυναμώσουμε. Αυτά ως σχόλια από πλευρά μου και προσβλέπω στην τελική έκθεση της κυρίας Ρούλε. Αυτά ως και εισηγητής λοιπόν ε, τη ομάδα μου και τώρα ω πρόεδρο να δώσω το λόγο στον κύριο Τριανταφυλλίδη να σχολιάσει από πλευρά του. Ε, ευχαριστώ κύριε πρόεδρε και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Ρούλε για την ε, πολύ ε, συλλογική προσέγγιση που έχει στο θέμα. Μας έδωσε την ευκαιρία σε συνάντηση που είχαμε μαζί της να εκφράσουμε τις απόψεις μας και θα έχουμε ακόμα μια συνάντηση αργότερα για να δούμε σε πιο, με πιο λεπτομερή τρόπο την όλη έκθεση. Θα ήθελα να κάνω κάποια συγκεκριμένα σχόλια. Ε, βλέπω μέσα από την έκθεση ότι τίθενται πάρα πολύ ορθά τα προβληματικά σημεία στις ε, δημόσιες συμβάσεις. Θα πρέπει να υπάρξει διασαφήνιση του κοινοτικού δικαίου ώστε να αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις του soft law που προέκυψαν από το δικαστήριο και προκαλούν νομική αβεβαιότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συντονίσει τη δράση της στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, ώστε να εκλείψει το φαινόμενο της διαφορετικής προσέγγισης από τα διάφορα τμήματα της Κομισιόν. Προβληματική είναι η συμπερίληψη περιβαλλοντικών, κοινωνικών ή άλλων ποιοτικών κριτηρίων στην αρχική περιγραφή του προϊόντος ή των υπηρεσιών που ζητούνται. Η έλλειψη σαφήνειας στις οδηγίες έχει δημιουργήσει την εντύπωση σε πολλούς ότι παρόλο που η καλύτερη αξία αποτελεί αποδεκτό κριτήριο, η χαμηλότερη τιμή είναι το μόνο κριτήριο που μπορεί να υποστηριχθεί με ασφάλεια. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη να γίνει πιο δυνατό το συγκεκριμένο σημείο στην έκθεση. Δεν αρκεί μόνο η αναφορά στην κοινωνική ευθύνη, αλλά θα πρέπει να γίνει αναφορά σε συγκεκριμένα μέτρα. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει και για τις περιπτώσεις των περιβαλλοντικών κριτηρίων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στην αγορά έτσι που να κατέχουν μερίδιο της ώστε με αυτόν τον τρόπο να επιβιώσουν. Θα πρέπει να προβάλλεται η σημασία της Δημόσιας Σύμβασης για τις μικρότερες επιχειρήσεις και να διευκολύνεται η πρόσβαση σε αυτές. Μως συνολικά πιστεύουμε ότι η εισηγήτρια έχει κάνει μια συνεχτική προσέγγιση επί του θέματος. Αναμένουμε ωστόσο να γίνει πιο ισχυρό το κείμενο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις αρμοδιότητες των περιφερειακών αρχών και για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Ευχαριστώ πολύ. Okay, well, I'd like to thank all the shadow Now... Ευχαριστούμε πολύ. Φαίνεται ότι το ενδιαφέρον είναι μεγάλο. Έχω 7 ε, ομιλητές. Μετά θέλω να δώσω το λόγο και στον εκπρόσωπο της Επιτροπής, αλλά και τελικά στην κυρία Ρούλο. Γι' αυτό σας παρακαλώ, έχουμε μισή ωρίτσα ακόμα, σας παρακαλώ να είστε σύντομοι. Θα σας δείχνουμε το ρολόι για να σας ε, ε, να φαίνεται ότι ο χρόνος πέφτει, φεύγει. Ωραία, λοιπόν, αυτοί είναι οι ομιλητές. Κλείνει ο κατάλογος. Χάνσεν πρώτος. Πρώτη μάλλον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας την εισηγήτρια η οποία ήρθε στο ύψος των περιστάσεων και των προκλήσεων Πρέπει να σας πω ότι εργάστηκα πάνω στο θέμα αυτό για μια άλλη επιτροπή ε, και πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει αρκετό συντονισμό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν ε, μιλάμε για τα διάφορα επιμέρους ζητήματα που άπτονται των δημοσίων ε, προμηθειών και συμβάσεων. Συγγνώμη. Επομένως, λείπει η απαραίτητη συνοχή, καθώς επίσης και ο συσχετισμός των κανονισμών της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις αφενός και τις διεθνείς συμφωνίες αφετέρου, οι οποίες όμως άπτονται και αυτές με κάποιο τρόπο των δημοσίων συμβάσεων. Το σημαντικό είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση των επιχειρήσεων της ευρωπαϊκή Ένωσης σε αυτές τις ε, συμβάσεις. Αυτό ε, αναφέρθηκε πολύ σήμερα. Η πρόσβαση λοιπόν αυτών των ευρωπαϊκών εταιριών σε τρίτες χώρες ε, και η δυνατότητα ελέγχου του ανταγωνισμού των επιχειρήσεων από τρίτες χώρες οι οποίες ε, θέλουν να ε, πάρουν δημόσιες συμβάσεις ε, στις χώρες μας. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν πολλές τρίτες χώρες οι οποίες έχουν κλειστή αγορά όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις τους και αυτό είναι κρίμα γιατί συνήθως ε, το αντίθετο συμβαίνει ε, από τη δική μας πλευρά. Δηλαδή οι εταιρείε από τρίτες χώρες έχουν πολύ πιο εύκολη πρόσβαση στις δικές μας δημόσιες ε, συμβάσεις. Αυτό θα πρέπει να το δει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι απαραίτητο να το ξαναδεί το θέμα έτσι ώστε να λειτουργήσουν καλά και όλες οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Α, ναι, δουλεύετε στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου για το θέμα αυτό. Έχετε δίκιο, ναι. Πολύ ωραία. Κυρία Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την κυρία Ρούλε για την εξαιρετική πρόταση. Είναι μια πολύ πλήρης ε, έκθεση, ε, γνωμοδότηση. Η πρώτη μου παρατήρηση είναι η εξής. Με την συνθήκη της Λισαβόνας έχουμε ένα νέο πρωτογενές πλαίσιο νόμου, ένα νομοθετικό πλαίσιο και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη απολύτως και πλήρως. Το θέμα της πολεοδομίας αναφέρθηκε ήδη διότι είναι εξαιρετικά σημαντικός. Βεβαίως, οι κοινότητες θέλουν να έχουν την ευχαίρεια να διαμορφώσουν το χωροταξικό τους περιβάλλον σε συνεργασία με τους πολίτες τους. Οπότε, έχει μεγάλη σημασία να διευκρινίσουμε ότι ένα σχετικό περιθώριο ελιγμών θα πρέπει να υπάρχει και να διασφαλιστεί Πρόκειται για τον ζωτικό χώρο, όχι μόνο για το οικονομικό περιβάλλον των πολιτών μας. Γι' αυτό είναι πολύ ε, απολύτως αναγκαίο να υπάρχει σαφήνεια σε όλες τις διατάξεις που αφαιρούν την πολεοδομία. Επίσης, όσον αφορά τώρα την ε, οδηγία ανάθεσης, ήμουν εισηγήτρια τότε όταν συζητούσαμε την οδηγία και θυμάμαι πολύ καλά τις διαβουλεύσεις. Είχαμε συζητήσει τότε εις βάθος εάν πρόκειται περί, του φθηνότερου, περί της φθηνότερης προσφοράς ή περί της βέλτιστης. Και το Κοινοβούλιο είχε αποφασίσει ότι θα πρέπει το βάρος, η ζυγαριά να γέρνει προς την βέλτιστη προσφορά την βέλτιστη προσφορά, την καλύτερη προσφορά από όλες τις απόψεις και όχι μόνο την φθηνότερη, την πιο οικονομική. Και γι' αυτό είχαμε πει ότι οι υπηρεσίες που κάνουν τον μειοδοτικό διαγωνισμό ε, θα πρέπει να λάβουν υπόψη και κοινωνικά κριτήρια και άλλα κριτήρια πέραν του κόστους. Αυτό είναι προφανές και έχουμε συμφωνήσει. Όμως διαπιστώνουμε ότι μεταξύ κομισιών και κρατών μελών υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες στην υλοποίηση αυτών των κριτηρίων, δηλαδή πώς θα καθορίσουμε τα κριτήρια και πώς θα εφαρμοστούν. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτό που είπατε κύριε Κρότσμαν, να αναθέσετε δηλαδή στην Κομισιόν την κατευθυντήρια γραμμή είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Επικίνδυνο κύριε Κρόιτσμα διότι δίνουμε την μονομερή εξουσία σε έναν φορέα. Ενώ εμείς πάντοτε ως κοινοβούλιο λέγαμε ότι οι δημόσιες ε, αυτές ε, αναθέσεις θα πρέπει να αποτελούν ένα μέσο που θα ωφελεί τις τοπικές αρχές, θα ωφελεί τις κοινότητες και που ενδεχομένως να αντιτίθεται στις ε, προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κομισιόν. Παρόλο που μπορεί να είναι αντίθετο, πρέπει να ωφελεί τις κοινότητες. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την κυρία Χάντσελ και τον κύριο Έγκελ. Πιστεύω ότι η έκθεση της κυρίας Ρίλε δεν έχω ακόμα την τελική έκθεση, η έχει ανασυνταχθεί, όπως είπε η συγγήτρια. Έχω μόνο την αρχική μορφή. Πάντως, είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η γνωμοδότηση και δεν θα μπορέσουμε δυστυχώς να ρυθμίσουμε πολλά σημεία έτσι όπως τα θέλουμε. Μία ανάθεση σε μία δημόσια σύμβαση είναι πάντοτε μία μεμονωμένη ανάθεση. Είναι μία περίπτωση, μία περίπτωση. Δεν μπορούμε λοιπόν σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση ανάθεσης δημόσιας σύμβασης να ανατρέχουμε σε συγκεκριμένη νομολογία. Η νομολογία και το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει για να καλύπτει γενικά το θέμα. Και γι' αυτό ακριβώς παρουσιάζονται και διαφορετικές ερμηνείες διότι σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση ανάθεσης προκύπτουν ερωτηματικά, προκύπτουν επικρίσεις, προκύπτουν διαφορετικές ερμηνείες. Άρα λοιπόν έχουμε αποφασίσει ότι θα πρέπει να ενισχύουμε τη βέλτιστη προσφορά. Αυτή να επιλέγεται και όχι η φθηνότερη. Βεβαίω τώρα διανύουμε μία εποχή με οικονομική στενότητα και δεσμεύσεις του προϋπολογισμού. Όμως πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο δεν θα προστατεύει αποκλειστικά τη φθηνότερη προσφορά. Εάν η Κομισιόν θέλει να προτείνει καινούργια ή συμπληρωματικά μέτρα, θα πρέπει να μας τα αιτιολογήσει σαφέστατα. εάν οι προτάσεις της προσβλέπουν στην διασαφήνιση νομικών ασαφιών, τότε ναι, είμαι διατεθειμένος να δεχτώ προτάσεις της Κομισιόν, αλλά μόνο εάν πρόκειται για ενίσχυση του πλαισίου και για διασαφήνιση ε, ασαφιών. Η κυρία Τέρνερ. Δεν ακούγεται. Πού Um, Ευχαριστώ πολύ. Σχετικά με τις ε, δημόσιες ε, συμβάσεις, πρέπει να πω ότι η έκθεση που έχουμε μπροστά μας είναι εξαιρετική. Για να μην ε, βαρύνουμε ακόμα περισσότερο τις τοπικές κυβερνήσεις με επιπλέον και τις τοπικές αρχές με επιπλέον γραφειοκρατικό άχθος θα πρέπει να έχουμε αρκετή ευελιξία. Δεν θέλουμε δηλαδή να δούμε τις ε, δημόσιες ε, συμβάσεις ε, με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τις δημόσιες προμήθειες. Νομίζω ότι οι προτάσεις της ηγήτριας είναι πολύ θετικές. Επίσης, ε, θα πρέπει πραγματικά να δούμε εάν είναι δυνατόν να περικόψουμε όσο γίνεται περισσότερο τις ανώφελες επιβαρύνσεις διοικητικές, γραφειοκρατικές κλπ έτσι ώστε να διευκολύνουμε όλους όσους εμπλέκονται σε αυτές τις δημόσιες συμβάσεις έτσι ώστε τελικά όλο αυτό το ζήτημα να αποβεί υπέρ των πολιτών. και βεβαίως η απάντηση, η σωστή απάντηση είναι οπουδήποτε υπάρχουν προβλήματα να ε, ε, προχωρήσουμε με περαιτέρω διασαφηνίσεις και να ανοίξουμε την αγορά, όχι να την κλείσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Η ε, κυρία Φερχάρη. Χωρίς μικρόφωνο. Δεν ακούν οι διερμηνείς. Καταρχάς, ευχαριστώ την κυρία Ρούλε από, από την πλευρά της Περιφερειακής Επιτροπής. Συνεργαστήκαμε θαυμάσια μαζί της. Είμαι σκιώδης εισηγήτρια για τη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Επιτροπής. Ήδη καλύφθηκα από τους ε, προλαλήσαντες. Αυτό το οποίο ζητήσαμε στην Περιφερειακή Επιτροπή είναι περισσότερη διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις, αλλά όχι απαραίτητο σε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο. Αυτή ήταν η γραμμή που υιοθετήσαμε. Και θέλω και επιμένω να τονίσω ξανά ότι χρειαζόμαστε μία πλούστευση των διαδικασιών, ιδίως για τις μικρές κοινότητες και για τις τοπικές αρχές, όπου είναι εξαιρετικά δύσκολο να ελεγχθεί και να πιστοποιηθεί η νομική ασφάλεια περίπλοκων συμβάσεων πολλές φορές έχουν δια... έχουμε διαπιστώσει ότι ευρωπαϊκές πιστώσεις δεν, διατέθηκαν σωστά, υπήρχαν ε, ατασθαλίες, αλλά λάθη θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί εάν υπήρχε απόλυτη σαφήνεια, μεγαλύτερη σαφήνεια και νομική ασφάλεια στην σύνταξη και δημοσίευση των μειοδοτικών διαγωνισμών. Πρέπει λοιπόν στις δημόσιες συμβάσεις να υπάρχει καλύτερη διαφάνεια έτσι ώστε να μπορούν επί του περιεχομένου να αξιολογήσουν την σύμβαση αυτή οι δημόσιες αρχές σε τοπικό επίπεδο, ακόμα και στο επίπεδο μιας μικρής κοινότητας. Πολλές φορές τα κείμενα είναι εξαιρετικά περίπλοκη. Επίσης, μια πλούστευση ε, της γραφειοκρατίας και της διατύπωσης θα ωφελήσει πολύ και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι πολλές από τις πιστώσεις αυτές, ε, ε, συγγνώμη, πολλές από τις συμβάσεις αυτές, ιδίως στον, κατασκευαστικό τομέα, δίνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και ακριβώ επειδή οι δημόσιε συμβάσει είναι τόσο περίπλοκε, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να αναλάβουν, δεν μπορούν να γίνουν ανάδοχοι. Σας ευχαριστούμε πολύ και είναι σημαντικό που έχουμε εδώ εκπρόσωπο και των, ε, της ε, Επιτροπής Περιφερειακών Υποθέσεων. Ευχαριστώ κυρία Τέρνερ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, δεν θα εκπλαγείτε εάν ε, σας πω ότι θεωρώ εξαιρετική την εργασία της κυρίας Ρούλη και αυτό δεν το λέω επειδή είμαστε στην ίδια πολιτική ομάδα, πρόκειται για μια πραγματικά εξαιρετική έκθεση γίνεται λόγος για λιγότερη γραφειοκρατία, γίνεται λόγος για ένα χτένισμα ε, των ε, ε, κανονισμών, των κανόνων, συγγνώμη, γιατί έχοντας ένα σωρό κανόνες και ένα σωρό διατάξεις τελικά δυσκολεύουμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο. Ε, βεβαίως ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο ε, να κινηθεί η τοπική διοίκηση σε αυτή την ζούγκλα. Χρειάζεται αποσαφήνιση, χρειάζεται σαφήνεια νόμου. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στις δύο μεγαλύτερες δανέζικες πόλεις οι αρχές αποφάσισαν ότι θα υπάρξει κοινωνική ρήτρα για όλες τις δημόσιες συμβάσεις. Ε, επομένως πρόκειται για ρήτρα η οποία διασφαλίζει, εγγυάται μάλλον την ε, κοινωνική διαστρωμάτωση ε, σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις. Όμως αυτό αντιτίθεται στην ουσία στον, στους υφιστάμενους ε, κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, όσον αφορά τις σχέσεις κεντρικής ε, και περιφερειακής αρχής και ξέρετε αρκεί να και αυτό έγινε στην περίπτωση της χώρας μου αρκεί κάποιος να έχει την ιδέα να δώσει μάχη όσον αφορά την ερμηνεία ενός υποκεφαλαίου που πραγματικά μπορεί να μπλοκάρει όλη την όλο το ζήτημα. Νομίζω ότι εδώ μας δίνεται πραγματικά η ευκαιρία να πάρουμε αποφάσεις οι οποίες θα διαφοροποιήσουν κατά πολύ το περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σουέκ. Ε, Ευχαριστώ. Σημείωσα το πρόβλημα. Είναι πρόβλημα πολυεθνικών καρτέλ κοινοπραξιών. Όταν μιλάμε για δημόσιες συμβάσεις πρέπει να σκεφτούμε την πραγματικότητα. Πώς εξελίσσεται όλη η διαδικασία. Οπωσδήποτε χρειαζόμαστε απλούστερους κανόνες. Αλλά εάν υιοθετήσουμε καινούργια στοιχεία, καινούργιες προτάσεις, πρέπει να έχουμε καλύτερο δημόσιο έλεγχο. Όταν πρόκειται για δημόσιες προμήθειες, η, μετά από έναν ε, διαγωνισμό θα πρέπει, να, θα πρέπει να δημοσιεύονται αυτοί οι ανάδοχοι, αυτοί που ανέλαβαν ε, τη σύμβαση και πληροφορίες για την εταιρεία τους, την επιχείρησή τους. Πρώτον λοιπόν διαφάνεια στην ενημέρωση. Δεύτερον, η διαφορά μεταξύ του, της συμφωνημένης ε, ε, σύμβασης, δηλαδή του ποσού της σύμβασης και του τελικού κόστους. Διότι πολλές φορές γίνεται ακριβώς μια τέτοια, ένας τέτοιος μειοδοτικός ε, ανταγωνισμός, ώστε λαμβάνουν την ανάθεση βεβαίως επειδή ήταν οι μειοδότες, αλλά συνεχεία τριπλασιάζεται ή πολλαπλασιάζεται το κόστος και πολλά από ε, τα κονδύλια αυτά είναι ευρωπαϊκά κονδύλια. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε αν υπάρχει υπερβολική και περίεργη διαφορά μεταξύ ανάθεσης και τελικού κόστους. Τρίτον, το διαφορετικό κατασκευαστικό κόστος ανάλογα με το έργο. Διαφορετικό κόστος έχει η κοινωνική κατοικία, διαφορετικό ένας αυτοκινητόδρομος. Πολλές φορές η διαφορά που υπάρχει στη, στην κοστολόγηση δεν είναι 5-10% είναι 200% και πολλοί μας κοροϊδεύουν ε, στην όλη διαδικασία δημοσίων συμβάσεων και δημοσίων διαγωνισμών ε, διότι ξέρουν ότι κάτι περίεργο κρύβεται από πίσω. Κάτι περίεργα πράγματα συμβαίνουν. Ο πρόεδρος πρέπει να δώσω το λόγο στην Κομισιόν αλλά δίνω το λόγο στον συνάδελφο για ένα λεπτό. Ε, συγχαίρω την εισηγήτρια και ιδίω ε, στο σημείο που αναφέρεται για τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Βεβαίως ε, θέλουμε να διασφαλίσουμε την ευελιξία και να μην ε, δεσμεύσουμε να μην στριμώξουμε υπερβολικά την εσωτερική αγορά. Εάν όμως κάνουμε παραχωρήσεις θα πρέπει να είναι σαφέστατα οριοθετημένοι. Έχουμε προβλήματα και στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Νόμου όσον αφορά την αποφυγή διακρίσεων, την ε, διαφάνεια. Όλοι είμαστε μπερδεμένοι. Υπάρχει μεγάλη σύγχυση. Άρα λοιπόν και χρειάζεται και σαφήνεια στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά καταφέρατε να είστε λακωνικός. Έχουμε τώρα τον εκπρόσωπο της Επιτροπής, ο οποίος θα μιλήσει δεν ξέρω αν θα μιλήσει και η κυρία Τσισκόφσκα, να δώσω από δύο λεπτά στον καθένα. Ξέρω ότι είναι πολύ λίγο το χρονικό διάστημα που σας διαθέτω, αλλά θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να το συζητήσουμε για να δώσουμε στη συνέχεια και το λόγο στην κυρία Ρούλη να συνοψίσει. Ενδεικτικό είναι το χρονοδιάγραμμα, αλλά σας παρακαλώ να είστε σύντομοι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Για την έκθεση και τα σχόλια που ακούσαμε σήμερα, νομίζω ότι μπορώ να πω ότι πολλές από τις ιδέες είναι κοινέ. Ε, ε, και οι δημόσιες προμήθειες έχουν δυνατότητες και για καλύτερη ε, εκμετάλλευση των πόρων μας αλλά και για καλύτερα έργα και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι στο οποίο συμφωνούμε όλοι. Το θέμα είναι πώς θα το επιτύχουμε. Όλα αυτά τα γνωρίζουμε, ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, ε, ελλείψεις σε πολλά θέματα και το θέμα είναι πώς μπορούμε να τα διορθώσουμε. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι μια ενδελεχή αξιολόγηση των κανόνων που έχουμε τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ε, να μην δώσουμε τόσο βάρος σε ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε εθνικό επίπεδο και από εκεί και πέρα ε, όσον αφορά στη σύνδεση με άλλες πολιτικές θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μιλά με μία φωνή. Δεν μπορούμε να έχουμε διαφορετικές γενικές διευθύνσεις να λένε διαφορετικά πράγματα. Ε, αυτό που είναι σημαντικό και το βλέπουμε και στην έκθεση είναι ότι θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι καταρχάς υπάρχουν δυνατότητες και νομίζω ότι αυτό αναφέρεται εν γέννη στην έκθεση και κατόπιν να αφήσουμε λίγο και ένα παράθυρο ανοιχτό σαφώς μπορεί να υπάρχουν και επικρίσεις ε, για το πώς θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε όλα αυτά που είδαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, όπως διαβάζουμε την έκθεση αυτή τη στιγμή είναι αρνητική ε, και είναι και αρνητική ως προς την αξιολόγηση που θέλουμε να κάνουμε. Νομίζω ότι είναι προς το συμφέρον όλων να πούμε ότι η πολιτική αυτή είναι σημαντική και οι δυνατότητες που υπάρχουν ε, θα πρέπει να ε, τις δούμε και να γίνει και με αξιολόγηση για να δούμε τι καλύτερη νομοθεσία ε, μπορούμε να έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ζητώ λοιπόν να είστε λίγο πιο ευέλικτοι στην έκθεσή σας. Ευχαριστώ η κυρία Τσισκόφσκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ίσως εντάχει και εγώ να πω δύο λόγια για ένα θέμα το οποίο είναι το θέμα των παραχωρήσεων δικαιωμάτων παροχής υπηρεσιών. Όσο έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει πάρα πολύ αναλυτικά όχι μόνο τι συμβαίνει στα κράτη-μέλη, αλλά και πολύ συγκεκριμένε περιπτώσει επιτόπου. Δεν υπάρχουν αποφάσει για τι διευκρινήσει που χρειαζόμαστε επί του θέματο αυτού. Επομένω, είμαστε ανοιχτοί προ συζήτηση και με τα κράτη-μέλη και με του ενδιαφερομένου. Θεωρούμε όμως ότι υπάρχει δυνατότητα να δράσουμε, υπάρχουν προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το θέμα είναι να εξεύρουμε τον καλύτερο τρόπο. Και ποια είναι τα προβλήματα, όπως ακούσαμε, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη έλλειψη διαφάνειας, δεν υπάρχει αντιμετώπιση ε, ισότιμη ε, σε επίπεδο κρατών μελών, δεν υπάρχει ισότιμο πεδίο για όλους, ε, δεν υπάρχει ε, καλή σχέση κόστου ωφελία και η αγορά είναι σχεδόν κλειστή για του εθνικού φορεί. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σα ε, στο γεγονό ότι οι παραχωρήσει δικαιωμάτων παροχή ή περιοχή είναι πολύ σημαντικέ όχι μόνο για την αξία του αλλά και για το γεγονό ότι διευρύνονται. Θα πρέπει λοιπόν, και αυτό προσπαθεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να βρει ένα πιο σταθερό και πιο λογικό τρόπο για να διεξάγονται αυτέ οι δραστηριότητε. Και οι λύσει είναι προ συζήτηση. Ευχαριστώ και τους δυο σας, λέει ο Πρόεδρος. Ε, είμαι βέβαιος ότι θα παρακολουθείτε το θέμα στενά και ε, σημειώνουμε τις παρατηρήσεις σας. Όπως είπα και εγώ, τα ωφέλη ε, αποτελεσματικών δημοσίων συμβάσεων είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει όλους. Να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Ρούλε για να συνοψίσει. Πριν όμως να σας πω λίγο το χρονοδιάγραμμα που προτείνεται, δεν ξέρω αν μπορείτε να με επιβεβαιώσετε και ότι εκρίνεται, προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών ε, επί του κειμένου σας 25 Μαρτίου, εξέταση τροπολογιών ε, στις 15 Απριλίου, ψηφίζουμε 28 Απριλίου στην Επιτροπή και περνάμε στην Ολομέλεια στο Μάιο. Αν ε, το δέχεστε θα μπορούσατε να μας το πείτε και επίσης να συνοψίσετε και για οτιδήποτε άλλο ακούσατε σήμερα το πρωί. Καταρχάς, ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη για τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους. Δεδομένου ότι ξέρουμε τις απόψεις των διαφορετικών ομάδων, θα είναι εύκολο να συγκεράσω αυτές τις απόψεις πριν από την ψηφοφορία. Σας είπα ότι έχω αλλάξει την δομή της γνωμοδότησης έχω διάφορα υποκεφάλαια, υποκεφάλαια, την έχω αναδιαρθρώσει και θα σας στείλω την τελική έκδοση. Έχω υιοθετήσει περισσότερα κοινωνικά ε, κριτήρια και έχω επίσης ένα καινούριο κεφάλαιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Και έχω διευκρινίσει καλύτερα τους γενικούς στόχους εκεί όπου ακόμα υπάρχει, υπάρχουν διαφορές με την Κομισιόν και εγώ και οι σκιώδεις ε, οι συγητές, είναι το, νομο, το νομοθετικό πλαίσιο και οι επιπτώσεις του. Λόγω της μεταφοράς του κοινοτικού δικαίου στα εθνικά δίκαια διαπιστώσαμε αυτές τις μεγάλες αποκλίσεις Αυτές οι αποκλίσεις έχουν δημιουργήσει μεταξύ ένα τεράστιο και περίπλοκο ε, ερμηνευτικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο δυσκολεύει αφάνταστα τη ζωή και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και των αναδόχων βεβαίως και όλων των ενδιαφεραμένων πλευρών. Γι' αυτό επιμένω ότι θα πρέπει να παγιώσουμε και να αξιολογήσουμε καταρχάς την υπάρχουσα νομοθεσία και εκεί χρειαζόμαστε την ενίσχυση και τη βοήθεια της Κομισιόν περισσότερο, όχι τόσο στην εκπόνηση νέων νομοθετικών μέτρων. Εγώ πιστεύω ότι η Κομισιόν θα πρέπει να συζητήσει τις κατευθυντήριες γραμμές Γι' αυτό υπάρχουν πολλές επικρίσεις, γι' αυτό το εγχειρίδιο ανάληψης κοινωνικής ευθύνης. Ε, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να επιβάλλουμε περισσότερη σαφήνεια, οπωσδήποτε περισσότερη σαφήνεια, όχι νέο νομοθετικό βάρος και ζητούμε να έχουμε όλα, όλη την τεκμηρίωση στα χέρια μας τουλάχιστον αυτή την οποία δίνει η Κομισιόν στα κράτη-μέλη. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Πολύ λίγα έγγραφα παίρνω εγώ στα χέρια μου. Άρα λοιπόν θέλουμε πλήρη ενημέρωση μέσω τεκμηρίωσης. Όσον αφορά τώρα τα concessions ε, και οι δύο οδηγίες ανάθεσης περιλαμβάνουν αιτιολογικό για αυτές τις... Ε, Zum τα, concessions, για αυτές τις παραχωρήσεις. Και ε, περιλαμβάνουν και συγκεκριμένη συγκεκριμένο ορισμό. Το Ευρωπαϊκό Δικοστήριο έχει υιοθετήσει, έχει αποδεχθεί αυτόν τον ορισμό των παραχωρήσεων. Μπορεί ορισμένα κριτήρια ακόμα να είναι αμφιλεγόμενα όσον αφορά ε, την διαφάνεια και την, τον καθορισμό των κριτηρίων για την παραχώρηση όμως οι ορισμοί έχουν δοθεί μέσω των δύο οδηγιών που ισχύουν. Ξέρω την γνώμη των κρατών μελών και τον οικονομικό τομέα. Κανένας δεν έχει διατυπώσει παράπονα για στρέβλωση του ανταγωνισμού και ο βιομηχανικός τομέας και ο κατασκευαστικός και οι τοπικές αρχές με, έκαναν έκκληση να μην επιβαρυνθούμε με περαιτέρω νομοθετικό βάρος. Προτού κάνουμε μία ολοκληρωμένη αξιολόγηση και παγίωση των ε, κανόνων της νομοθεσίας. Υπάρχει τέτοια μεγάλη πληθώρα κανονισμών και νόμων που πρώτα πρέπει να, να χωνευτούν, να παγιωθούν και μετά να έχουμε καινούριου. Πρόεδρος, να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετέσχουν σε αυτήν την πάρα πολύ επικοδομητική συζήτηση. Πολλοί ζήτησαν το λόγο και αυτό από μόνο του δείχνει το ενδιαφέρον που αποδίδουμε ε, στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστούμε όλους που πήρατε το λόγο για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Ωραία και το χρονοδιάγραμμα από ό,τι κατάλαβα δεν σας δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Επομένως, προχωράμε στο τελευταίο σημείο για σήμερα το πρωί. Έχουμε 15 λεπτά. Ε, για να συζητήσουμε για το θέμα της βελτίωσης της λειτουργίας αλυσίδας ε, τροφίμων στην Ευρώπη. Αποφασίσαμε, επιλέξαμε δηλαδή να κάνουμε γνωμοδότηση για το θέμα αυτό. Ο κύριος Φόξ θα ε, εκπονήσει την έκθεση. Είναι εδώ για να ανταλλάξει κάποιες απόψεις μαζί μας. Έχουμε επίσης ε, τον κύριο Ζουβά, ο κύριος Μπεζόη νομίζω ότι θέλει να μιλήσει. Ξέρω με τον κύριο Λάιον που απουσιάζει. Δεν ξέρω αν οι πράσινοι θα μιλήσουν αλλά εάν κάποιος θέλει από τους πρασίνους να συμβάλλει στη συζήτηση. Λοιπόν, επίσης να παρακαλέσω τους αποχωρούντες να αποχωρήσουν ισχύος Και να δώσω αμέσως το λόγο στον κύριο Φόξ για να μας πει τι σκοπούς έχει για αυτή τη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όσοι είδαν την έκθεση Μποβέ θα έχετε ε, καταλάβει ότι το πεδίο είναι εξαιρετικά ευρύ. Εγώ σκοπεύω να αναφερθώ στη γνωμοδότηση μονάχα στα θέματα της εσωτερικής αγοράς και προστασίας του, ε, των καταναλωτών έτσι ώστε να ε, συρρυκνώσω λίγο το πεδίο που ήταν πολύ ευρύ και πολύ φιλόδοξο από τον κύριο ε, Βοβέ. Πιστεύω ότι 7 από τις συστάσεις είναι ε, ιδιαίτερα σημαντικό, ε, σημαντικά για την Επιτροπή μας. Ε, δεύτερον, πρώτο θέμα, η έλλειψη άρσης τρέβλωσης του ανταγωνισμού. Δεύτερον, η ευκολία πρόσβασης στο αναλώσιμα της αγοράς. Τρίτον, εργαλεία εποπτείας και στατιστικής. Τέταρτον, σύσταση ε, προς όλα τα κράτη-μέλη να έχουν παρατηρητήρια τιμών και υπηρεσίες ε, οι οποίες θα ασχολούνται με σύγκριση τιμών λιανικής ε, στο διαδίκτυο επίσης έλεγχο των, των μεγάλων διαφορών των τιμών, επίσης θέματα που σχετίζονται με την σήμανση των προϊόντων, τις ετικέτες κλπ. Ε, και τέλος το θέμα το οποίο σχετίζεται με, την προστασία των καταναλωτών όσον αφορά την πιστοποίηση ε, των ε, ουσιών που είναι επικίνδυνες για την ουσία. With και η καταγραφή τους στη σήμανση των προϊόντων είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει μια σωστή ε, αλυσίδα ε, διατροφής ε, η οποία θα διατηρεί συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων. Πιστεύω ότι ο στόχος μας θα πρέπει να είναι καταναλωτές όλο και πιο καλά ενημερωμένοι και η σωστή εποπτεία της αγοράς θα βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου αυτού. Όσον αφορά την εσωτερική αγορά, φαίνεται ότι υπάρχουν διαφορές στην δυνατότητα διαπραγμάτευσης που έχουν διάφορες ομάδες. Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι η ελεύθερη αγορά μπορεί να λειτουργήσει ε, όταν ε, οι επιδοτήσεις ε, δίνονται με σωστό τρόπο τότε έχουν ως αποτέλεσμα καλής ποιότητας προϊόντα στην διάθεση των καταναλωτών αγοραστών. Αλλά για να λειτουργήσει καλά όλο αυτό το σύστημα τότε θα πρέπει να υπάρξει διαφάνεια αφενός και ξεκαθάρισμα κατά κάποιο τρόπο της αγοράς από τους μεγάλους υπερβολικά σημαντικούς παίκτες. Πιστεύουμε ότι ε, θα πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί η δεσπόζουσα θέση ε, κάποιων ε, ενδιαφερόμενων και εμπλεκόμενων στην αγορά. Ε, γιατί σε αυτήν την περίπτωση στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός και τα προϊόντα που φτάνουν στην αγορά και τελικά στον καταναλωτή δεν φτάνουν με τους καλύτερους δυνατούς τρόπους. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει ε, εισαχθεί ένας νέος κώδικας ε, ο οποίος βεβαίως θα πρέπει να ελεγχθεί ως προς την αποτελεσματικότητά του. Καλωσορίζω την ε, σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, όσον αφορά ε, τον κατάλογο βελτίστων πρακτικών και συμμερίζομαι την ανάγκη να υπάρχει ένας τέτοιος κατάλογος κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι η επιλογή μου να αναφερθώ μονάχα σε θέματα εσωτερικής αγοράς και προστασίας καταναλωτών θα αποβεί τελικά υπέρ της γνωμοδότησης, γιατί θεωρώ ότι ε, ακριβώς μειώνοντας ε, το πεδίο εφαρμογής μπορούμε να έχουμε πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Πρόεδρος, ναι, είναι αλήθεια. Ε, αναφερθήκατε σε 7 τομείς προτεραιότητας ε, που είναι πάρα πολύ σημαντικοί και νομίζω ότι έχετε τη σωστή προσέγγιση. Ο κύριος Ζουβέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούστε με, Πρόεδρε. Ε, είναι εξαιρετικά διαφωτιστική η ανάγνωση της έκθεσης Μποβέ της οποίας συμμερίζομαι όλα τα θέματα και όλα τα ζητήματα. Γιατί για να δούμε πώς έχει η κατάσταση. Πριν από μερικά χρόνια, το 1960, οι χώρες ε, της ΕΟΚ τότε είχαν ε, μία αυτάρκεια τροφίμων της τάξης του 80%. Δημιουργείται η ΚΑΠ, η αυτάρκεια φτάνει στο 100% μετά από 10 χρόνια αλλά λίγο μετά αρχίζει να χαλάει το σύστημα με τα τεράστια αποθέματα τα οποία γνωρίζουμε όλοι που στρέβλωσαν τελικά το ε, σύστημα. Και βεβαίω το θέμα των ποσοστώσεων στο γαλακτοκομικό τομέα νομίζω ότι είναι διαφορετικό για όλους. Γνωρίζετε επίσης ότι η Ευρώπη είναι και καθαρός εξαγωγέας. Λαμβάνοντας λοιπόν όλα τα ζητήματα αυτά υπόψη, εάν υποτιμήσουμε τα όσα αναφέρει ο κ. Μποβέ, ενδεχομένως θα φτάσουμε στο μέλλον σε μια κατάσταση όπου η αυτάρκεια τροφίμων ε, δεν ε, θα είναι δεδομένη. Βεβαίως ε, κατανοώ ότι μερικοί λένε ότι η αυτάρκεια των τροφίμων δεν είναι αυτός σκοπός, αλλά αλλά αυτή η ιστορική στάση ε, τελικά αναθεωρήθηκε όταν οι τιμές των πρώτων υλών πριν από μερικά χρόνια ε, ε, αυξήθηκαν αστρονομικά και έφτασαν στα αστρονομικά επίπεδα. Και αυτό μπορεί να συμβεί και στο μέλλον. Δεν κατανοούμε τελικά το μηχανισμό, δεν κατανοούμε γιατί οι τιμές ανεβαίνουν για τους καταναλωτές αλλά τελικά δεν καρπούνται την ε, αύξηση αυτή η παραγωγή ε, και επομένως κατανοούμε ότι το σύστημα των επιδοτήσεων τελικά με κάποιο τρόπο δεν λειτουργεί καλά. Ε, και Επομένως δημιουργούμε κάποια επιπλέον εθνικά εργαλεία, παρατηρητήρια όπως τη Γαλλία ας πούμε έτσι ώστε να προσπαθήσουμε καλύτερα να κατανοήσουμε τα προβλήματα αυτά γιατί είναι γεγονός ότι εμφανίστηκαν κάποιοι νέοι εμπλεκόμενοι, τους οποίους δεν γνωρίζαμε. Στη Γαλλία 20% των γευμάτων ε, καλύπτονται από τους ε, βιομήχανους που ασχολούνται με τη μαζική εστίαση. Και δεν καταλαβαίνουμε τελικά πώς λειτουργούν πλέον οι διατροφικές αλυσίδες. Επομένως, πριν πάρουμε οποιαδήποτε απόφαση, ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε καλύτερα τι συμβαίνει. Ας προσπαθήσουμε να δούμε καλύτερα ε, για ποιο περιβάλλον μιλάμε. Όπως είπα και στην αρχή της παρέμβασής μου, συμφωνώ με όλα αυτά που λέει ο κύριος Μποβέ στην ε, έκθεσή του. Α, τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να σκεφτούμε όλοι μαζί έτσι ώστε να θέσουμε τα σωστά ερωτήματα έτσι ώστε να μην δυναμητιστεί η δυνατότητα της Ευρώπης να έχει διατροφική αυτάρκεια. Όλα αυτά τα θέματα είναι και θέματα εσωτερικής αγοράς, κύριε Φόξ, και θα συμφωνήσω μαζί σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τη συνεργασία με τον εισηγητή κύριο Φόξ και τους άλλους σκιώδης εισηγητές. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική έκθεση για όλους τους καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι θα επιβάλλει μια ε, σαφήνεια για την όλη αλυσίδα ε, εφοδιασμού και διανομής ε, των τροφίμων, τις διαφορές των τιμών, Υπάρχει πραγματικά μια μεγάλη ανισορροπία στις τιμές που διατίθενται τα προϊόντα και στις τιμές που λαμβάνουν οι παραγωγοί. Θα ήθελα να ε, κάνω μερικές παρατηρήσεις όμως. Οι παραγωγοί δεν παράγουν μόνο προϊόντα, αλλά σήμερα είναι και μεσάζοντες πολλές φορές. Δεν είναι λοιπόν μόνο η, αρχή της αλυσίδας, αλλά αποτελούν και κρίκο στο μέσο της αλυσίδας. Αυτή λοιπόν η, αλλαγή των δραστηριοτήτων τους πρέπει να φωτιστεί, πρέπει να αποσαφινιστεί περαιτέρω. Η Κομισιόν έχει ένα πρόβλημα. Εφόσον δεν υπάρχουν αποδείξεις για στρεβλώσεις της αγοράς, η αγορά είναι ελεύθερη να δράσει ανεξέλεγκτα. Ξέρουμε ότι πάρα πολλές ε, συμφωνίες κλείνονται χωρίς ε, να υπάρχει γραπτή απόδειξη, γραπτή σύμβαση. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα αλεξέλεγκτο στοιχείο. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχουν αποδείξεις, δεν μπορούν να υπάρχουν και προσφυγές στα δικαστήρια σε περίπτωση παρανομιών ή στρεβλώσεων της αγοράς. Πολλές φορές αυτός ο οποίος αγοράζει την πρώτη ύλη, ο παραγωγός ε, δηλαδή και εν συνεχεία μετατρέπεται σε μεσάζοντα για να πουλήσει τα προϊόντα του, αναγκάζονται από τον κατασκευαστή της πρώτης ύλη να σιωπήσουν, δηλαδή να αποκρύψουν τις πρώτες του ύλε και τις πηγές εφοδιασμού, τις πηγές προμήθειας για διάφορους λόγους. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα στους παραγωγούς να εξαλειφθεί αυτή η στρέβλωση, αυτή η παραβίαση των κανόνων έτσι ώστε όλες οι πηγές προμήθειας και των πρώτων υλών αλλά και εν συνεχεία οι επόμενες φάσεις στην ε, ε, τροφική παραγωγή να είναι ξεκάθαρες και σαφείς. Εάν υπάρχουν στεγανά και αν υπάρχουν κρυφές πτυχές, αυτό διακινδυνεύει την ποιότητα των τροφίμων για τους καταναλωτές. Θα πρέπει λοιπόν να καταπολεμήσουμε τέτοιες ε, κρυφές ή μυστικές διαδικασίες. Γι' αυτό χαίρομαι που θα συνεργαστώ με τον εισηγητή και τους άλλους και όδης Θα, είμαι σίγουρη ότι θα υπάρχει μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση η οποία θα διευκρινίσει πολλές απορίες που υπάρχουν. Ευχαριστώ ο κύριος Μπουζόη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς ο κύριος Λάνος, ο σκιώδης συγητής, είναι στην Επιτροπή Γεωργίας διότι έχουν προγραμματιστεί ψηφοφορίες ταυτόχρονα αλλά συζήτησα μαζί του και θα ήθελα να σταθώ σε τρία σημεία εκ μέρους του και εξ ονόματος της αντιπροσωπείας μας εδώ. Πρώτον, θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη να ενισχυθούν ε, οι δυνατότητες διαπραγμάτευσης των προμηθευτών σε σχέση με τους παραγωγούς ε, οι οργανώσεις παραγωγών έχουν να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο στο θέμα αυτό. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αντιεμπορικές πρακτικές και όχι μόνο να ανταλλάσσουμε πληροφορίες για τις πρακτικές αυτές και θα πρέπει να δούμε και την πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή βέβαια δεν προτείνουμε να δούμε το σύνολο της πολιτικής ανταγωνισμού αλλά φρονούμε ότι θα πρέπει να κάνουμε κάποιες μικροδιορθώσεις προκειμένου να ενισχύσουμε τις θέσεις των αγροτών. Δεύτερον, Είμαστε υπέρ της ε, ε, τάσης για μεγαλύτερη διαφάνεια, θέλουμε να συλλέγονται περισσότερα δεδομένα για τις τιμές, αλλά όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται από ανεξάρτητο φορέα και όχι απαραίτητα από τον ίδιο τον τομέα. Και εδώ τίθεται και το ερώτημα τι ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν τα μέσα ευρωπαϊκής παρακολούθησης των τιμών θα πρέπει να υπάρχει και κάποιο ε, διαμεσολαβητής, κάποιος ombudsman για να εξετάζει τι γίνεται με θέματα τιμών. Η Γερμανία έχει ήδη συμφωνήσει στο να υπάρχει κάποιο αντίστοιχος ε, ε, διαμεσολαβητής και ίσως θα πρέπει να έχουμε και κάποιον σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να δούμε και τι εξουσίε θα πρέπει να έχει ο διαμεσολαβητή. Είμαστε βέβαιοι ότι οι συζητήσεις εδώ στην Επιτροπή μας ε, και η γνωμοδότηση η οποία θα προκύψει από, τον, ε, από τη συζήτηση και τη οποία συντάκτη είναι ο αξιότιμο κύριος Φόξ, θα ενισχύσει τη θέση των εργατών και θα μα βοηθήσει ε, στα θέματα τη Επιτροπή Γεωργία, η οποία είναι και η αρμόδια επί τη ουσία επιτροπή για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ κύριε Μπουσόη. κύριε Ρούλε. Θα είμαι πολύ σύντομη γιατί καλύφθηκα από τους προλαλήσαντες. Ευχαριστώ τον κύριο Φόξ Σίγουρα η γνωμοδότηση αυτή θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα και πιστεύω ότι και στις ομάδες υπάρχει συνένεση. Όσον αφορά τώρα τις γεωργικές επιδοτήσεις, όταν συζητούσαμε τη διαφάνεια, είπαμε ότι επιδοτήσεις που δίδονται από το κράτος πηγαίνουν σε εταιρείες κατασκευής, ε, παρασκευής τροφίμων. Οπότε εκεί ενδέχεται να σημειώνεται στρέβλωση της αγοράς. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Αν πηγαίνουν επιδοτήσεις ε, επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων. Δεύτερη παρατήρηση, συγκέντρωση της αγοράς, καρτέλ, ε, δεσπόζουσα θέση δηλαδή ενός καρτέλ μιας κοινοπραξίας. Αυτή η πτυχή δεν έχει εξεταστεί επαρκώς. Πρέπει να εξετάσουμε τι γίνεται στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Διότι στα τρόφιμα έχουμε ήδη μια πολύ υψηλή συγκέντρωση επιχειρήσεων, σύμπραξη επιχειρήσεων. Κίνδυνος λοιπόν πολύ ισχυρών καρτέλ. Οπότε τίθενται πολλά ερωτήματα, μήπως πηγαίνουμε προς την κατεύθυνση ε, μονοπωλίων ε, ε, Ιδίω στον γαλακτοκομικό τομέα που γίνονται πολύ σκληρέ διαπραγματεύσει. Μήπως εφαρμόζεται το δίκαιο των κοινοπραξιών μονόπλευρα προς όφελος της μίας πλευράς των επιχειρήσεων και όχι των παραγωγών. Εξπεραιτέρω εξέταση λοιπόν αυτού του ζητήματος και υποστηρίζω τις βέλτιστες πρακτικές, best practice, όλα τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ πολύ δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Ξέρω ότι έχουμε κάποιον εκπρόσωπο της Επιτροπής εδώ. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιες σύντομες παρατηρήσεις, να πείτε και λίγα λόγια για εσάς στην Επιτροπή και είμαι σίγουρος ότι θα σας ξαναπροσκαλέσουμε για να συζητήσουμε για το θέμα αυτό. Αν θέλετε σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Πιέρ Λουίτζι Λοντέρο λέγομαι, εργάζομαι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Ανάπτυξης Πέθρου. Ήμουν υπεύθυνο μαζί με άλλους συναδέλφους ε, από άλλες αρμόδιες γενικές διευθύνσεις, 8 για την ακρίβεια, για την εκπόνηση της ανακοίνησης για την καλύτερη λειτουργία της ε, αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμου. Εχθές έγινε μια πρώτη συζήτηση στην Γενική Διεύθυνση Γεωργίας για το έγγραφο εργασίας που ετοίμασε ο κύριος Μποβέ. Είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ φιλόδοξο έγγραφο εργασίας, το οποίο θα οδηγήσει, φαντάζομαι, και σε μία ανάλογα φιλόδοξη έκθεση. Από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεωρούμε ότι ο κατάλογος των θεμάτων και επισημάνσεις των αδυναμιών της ανακοίνωσης μάλλον υπερβαίνει το πεδίο εφαρμογής ανακοίνωσης. Η ανακοίνωση ε, ήταν ουσιαστικά μία συνέχεια των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία παρακολουθούσε το κατά πόσον λειτουργούσε καλά η αγορά ε, κατά το διάρκεια του 2007 και 2008 όσον αφορά στις τιμές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στάθηκε σε δύο σημεία που είναι ο μηχανισμός διαβίβασης των τιμών και ε, τα στατιστικά στοιχεία για τις τιμές ε, και έγιναν και κάποιες συστάσεις από αυτού. Η έκθεση του κυρίου Μποβέ ε, είναι πολύ πέραν αυτών των θεμάτων και θεωρούμε ότι θα ήταν ένα καλό μέσο για να ξεκινήσουμε μια συζήτηση η οποία ελπίζουμε να αποβεί καρποφόρα. Εχθέ ε, ήρθαμε σε επαφή και με τον κύριο Φόξ ε, για τη δική του τη γνωμοδότηση και ε, είμαστε καθόλου πρόθυμοι για συνεργασία. Με αυτά νομίζω ότι αρκεί. Θα δώσω σχόλια στον εισηγητή, τον κύριο Μποβέ, για τα στοιχεία τα οποία επισημαίνει στην έκθεσή του και θα επανέλθουμε φυσικά στο θέμα αυτό και στη δική σας την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί σας. Κύριε Φόξ, μήπως θέλετε να συνοψίσετε, να προτείνω και ένα χρονοδιάγραμμα, να δω κατά πόσον το δέχεστε, ε, το οποίο συνάδει και με τα όσα κάνει η Αρμόδια Επιτροπή. Θα αποστείλετε το κείμενό σας για μετάφραση μέχρι τις 8 Απριλίου. Θα εξετάσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης ε, πιο διεξοδικά 22 και 23 Απριλίου. Θέλουμε να έχουμε αρκετό χρόνο γιατί φαντάζομαι ότι θα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ε, κατάθεση τροπολογιών μέχρι τις 10 Μαΐου, εξέταση των τροπολογιών 2 Ιουνίου και ψηφοφορία στις 3 Ιουνίου στην Επιτροπή μας και κατόπιν η αρμόδια θα ψηφίσει 8 ε, Ιουνίου η αρμόδια Επιτροπή. Φαντάζομαι ότι αυτό θα σας δώσει και το χρόνο να διαπραγματευτείτε μαζί σας για να περάσουν οι απόψεις της Επιτροπής μας. Ε, αν θέλετε να συνοψίσετε λοιπόν και να μου επιβεβαιώσετε και κατά πόσον δέχεστε το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Απολύτως αποδεκτό το χρονοδιάγραμμα. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω όσα είπαν οι συνάδελφοι. Του ευχαριστώ για τη συνεισφορά του και ε, προσβλέπω στη συνεργασία με όλου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λίγη τη συνεδρίαση. Σας παρακαλώ να έρθετε στις 3 ακριβώς, ε, γιατί έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τον Ισπανό Υπουργό στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να συζητήσουμε όλα τα θέματα που αφορούν την Επιτροπή μας, καθώς επίσης και στόχους για τη στρατηγική του 2020. Ε, θα ήθελα να είστε όλοι παρόντες εδώ. Καλή όρεξη και θα επανέλθουμε Δημήτρη στις 3.